Dear colleagues, Λοιπόν, ε, να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας ε, με το σημείο 11, ανταλλαγή απόψεων για την Μέση Ανατολή και την ειρηνευτική διαδικασία. Καλωσορίζουμε τον κύριο Τζεντιλίνη, τον ειδικό εκπρόσωπο των Ηνωμένων για την, ε, για την ειρηνευτική διαδικασία των Μέσων Εθνών, μαζί με τον πρέσβη Πιέρ που το ξέρουμε. Και τώρα είναι ο ειδικό απεσταλμένο του Υπουργείου Εξωτερικών τη Γαλλία για το ίδιο θέμα. Και τον δόκτωρα Αρμάν Μπένμια που είναι καθηγητή διεθνών σχέσεων και μέσα ανατολικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Όλοι αυτοί ε, γνωρίζουν ιδιαίτερα το θέμα και ελπίζουμε η τελευταία αποτίμηση της κατάστασης έγινε τον περασμένο Ιούλιο και η ομάδα εργασίας, το κουαρτέτο, ε, όρισε τρία κυρίως προβλήματα για την ειρηνευτική διαδικασία. Η, βία στην Παλαιστίνη, η επέκταση των οικισμών σε περιοχές που έχει σημειωθεί για να ε, ε, ανήκει στο Παλαιστινιακό κράτος και η, ο, η, η έλλειψη ελέγχου της Παλαιστινικής Αρχής στη Γάζα. Τι συνέχισε έχει δοθεί σε αυτά τα τρία θέματα, τι συνέχισε έχει δοθεί σε αυτή την έκθεση του κουαρτέτου, ποιε είναι οι πρόσφατες εξελίξεις, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, πολύ καλή ευκαιρία είναι αυτή μαζί με τον Πιέρ Βημό να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Σε αυτήν ακριβώς τη φάση. να εστιάσω σε τρία κυρίω σημεία. Υπάρχουν και πολλά άλλα, αλλά αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Και μετά ίσως να αναφερθώ και στα άλλα. Κατά την ανταλλαγή απόψεων. Καταρχάς, θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο από πριν στην ε, λύση μέσω δύο κρατών. Να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε, δηλαδή αυτή τη δυνατότητα αυτό το κεκτημένο. Και μετά θα ασχοληθώ με τις διάφορες ε, πρωτοβουλίες για να επιτύχουμε αυτή τη λύση. Αναφερθήκατε στην έκθεση του κουαρτέτου κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι και ο Πιέρ θα μας πει κάτι για τη γαλλική πρωτοβουλία. Και μετά να αναφερθώ σε αυτά που ήδη κάνετε και τι μπορείτε κι εσείς να κάνετε περαιτέρω για να συμβάλλετε. Λοιπόν, λύση μέσω δύο κρατών. Αυτή είναι η θέση, η σαφή θέση της Ένωσης. Είναι μια θέση που την ε, αναγνωρίζουν και οι δύο πλευρές και στηρίζεται από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Μοιάζει να είναι προφανής λύση, αλλά αυτό το προφανές δεν είναι τόσο προφανές σε αυτή τη συγκυρία. Σε αυτή τη συγκυρία πρέπει πραγματικά να το διατηρήσουμε αυτό. Οι τάσεις και η δυναμική σε αυτή τη συγκυρία δεν είναι ενθαρρυντικές. Λόγω διαφόρων στοιχείων. Υπάρχει ε, ουσιώδης έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Ε, κάποια γεγονότα για την συνεργασία για την ασφάλεια, για άλλες πρωτοβουλίες, μια πρωτοβουλία συμφωνίας για την ενέργεια. Αλλά ε, παρόλα αυτά οι δύο πλευρές δεν έχουν ε, επιτύχει να επανέλθουν σε ουσιώδεις συζητήσεις και Κάποια γεγονότα επιτόπου δεν βοηθούν. Για παράδειγμα, η παρέμβαση, όπως είπε πριν από μια εβδομάδα η Φεντερίκα Μογκερίνη στην Ολομέλεια, όπου ακριβώς περιέγραψε την κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Την περιέγραψε αναλυτικά και έγινε και ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχουν και ε, προβλήματα και περιορισμοί εσωτερικής πολιτικής και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, πρέπει να ασχοληθούν και με άλλα θέματα. Ξέρουμε πολύ καλά πώς έχει η κατάσταση στο Ισραήλ, ε, τι περιθώρια δράσεις υπάρχουν προς τη λύση των δύο κρατών λόγω του υπάρχοντος συνασπισμού στην κυβέρνηση του Ισραήλ και στην Ραμάλα. Υπάρχει πολύ ένταση για εσωτερικά θέματα. Σήμερα είχαμε την ε, διάσκεψη της ε, ΦΑΤΑ, σήμερα ξεκινάει, να δούμε πού θα καταλήξει, αν θα αποσαφινιστεί η κατάσταση. Αλλά τα θέματα αυτά οπωσδήποτε είναι σημαντικά. Υπάρχουν και άλλα πολύ πιεστικά θέματα στην περιοχή. Νέα Αμερικανική κυβέρνηση που θα αναλάβει σε λίγο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Οι περιστάσεις. Και γι' αυτό τονίζω περισσότερο παραποτέ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η λύση των δύο κρατών είναι αυτή που θέλουμε να προωθήσουμε και δεν υπάρχουν ρεαλιστικές αναλλακτικές. Χθες συναντήθηκα με μερικούς νέους ε, Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους ηγέτες, νεαρούς δηλαδή. Ήταν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Φυσικά οι άνθρωποι ε, πέφτουν σε όλο και περισσότερη απόγνωση όσο βλέπουν πως δεν προωθείται τίποτα. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να πιέσουμε, να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε το ρεύμα. Όπως ακριβώς το είπε και το κουαρτέτο, η βία, η εξώθηση σε βία, οι οικισμοί και η Γάζα. Για να αποκτήσουν ε, οι πολίτες της Επιτόπου ε, κάποια ελπίδα μέσω και βελτίωσης των ε, συνθηκών ζωής τους. Προσπαθούμε. Με ρωτήσατε τι συνέχιση υπάρχει, τι συνέχεια έχει δοθεί στην έκθεση. Αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε να συνεχιστεί να υπάρχει εστίαση και ενότητα της διεθνούς κοινότητας, ούτως ώστε οι προτάσεις για να αποκτήσουν ε, περισσότερες αρμοδιότητες οι Παλαιστίνοι στα πλαίσια των περιορισμών ασφαλείας, να προθεθούν με κάποιο τρόπο όλα αυτά. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε σε αυτήν τη συγκυρία. Είναι σημαντικό το ότι υπήρξε έκθεση του κουαρτέτου, γιατί είναι μια κοινή αποτίμηση της κατάστασης από τους κύριους ε, πρωταγωνιστές, Ηνωμένα Έθνη, Ηνωμένε Πολιτείες, Ρωσία, Ένωση. Περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό δεν είναι αμεληταίο. Θέλουμε να γίνουν, τα βήματα που θέλουμε να γίνουν είναι πραγματική αλλαγή της κατάστασης. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερες εξουσίες στους Παλαιστινίους, λαμβάνοντας υπόψη τις νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας του Ισραήλ. Αλλά σε τελευταία ανάλυση μπορούμε να πιέσουμε, μπορούμε να επιχειρήσουμε να ενθαρρύνουμε, μπορούμε να συστήσουμε μηχανισμούς για να προωθηθούν όλα αυτά, αλλά σε τελευταία ανάλυση ε, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση των δύο πλευρών. Αυτό είναι το πραγματικό θέμα, διότι οι προτάσεις που παρουσιάσαμε δεν είναι και τόσο καινούργιες. Όποιος γνωρίζει την κατάσταση ξέρει ότι οι προτάσεις και από τις δύο πλευρές είναι περίπου ίδιες αυτών που ενδιαφέρονται για την ειρήνη. Άρα το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, να πιστούν δηλαδή ότι είναι καλό και για τις δύο πλευρές να υπάρξει αυτή η λύση. Γι' αυτό παίζει ρόλο να υπάρχει ενιαία στάση του διεθνούς παράγοντα, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη. Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει καμία αξιόπιστη εναλλακτική. Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα, αλλά αν και όποτε θέτω το ερώτημα τι άλλη λύση θα ήταν ρεαλιστική, δεν έχω λάβει πιστικές απαντήσεις. Θέλουμε ένα δημοκρατικό εβραϊκό Ισραήλ, θέλουμε ένα κράτος για τους Παλαιστινίους που είναι οι νόμιμες διεκδικήσεις τους. Αν θέλουμε να απαντήσουμε ναι, όπως πιστεύω ότι θα έπρεπε να απαντήσουμε και, σε αυτές τις, και στις δύο αυτές ερωτήσεις, δεν βλέπω άλλη εναλλακτική. Πρέπει να βαδίσουμε προς αυτή την λύση των δύο κρατών. Μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλειών εν εξελίξη μίλησα για το κουαρτέτο, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι κυρίως πρέπει να εστιάσουμε στην ίδια την ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει αραβική πρωτοβουλία για την ειρήνη. Εκεί είναι και για τις δύο πλευρές τα πραγματικά κίνητρα για να βαδίσουν προς αυτή τη λύση. Πρέπει λοιπόν να εμπλακεί η περιοχή ευρύτερη. Αυτό προσπαθώ να κάνω, συμβάλλοντας ε, στην ε, δουλειά της Ένωσης γι' αυτό, διότι αν υπάρξει μια πρωτοβουλία, μια πρόταση από τις χώρες της περιοχής, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική από μια πρόταση από άλλο μέρος του κόσμου. Είμαι σε μόνιμη επαφή με τους Αιγύπτιους, τους Ιορδανού, τους Σαουδάραβες, τον Αραβικό Σύνδεσμο. Είναι σημαντικό να υπάρξει πρόοδος από αυτού. Δεν ε, νομίζω ότι αγνοούμε τις άλλες προκλήσεις που έχουμε στην περιοχή. Δεν είναι ότι έχουμε αποκλειστικά επικεντρωθεί σε αυτήν την ιδέα και δεν ξεχνάμε τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά υπάρχουν και άλλες πιεστικές προκλήσεις στην περιοχή. Αλλά η πρόοδος στο ισραλο παλαιστινιακο θα αφαιρέσει ένα από τα κύρια αίτια της ριζοσπαστικοποίησης της περιοχής και θα ξεμπλοκάρει και άλλε δυνατότητε επίλυση άλλων προβλημάτων στην περιοχή. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να θέτουμε έτσι το θέμα προ όλε τι πλευρέ. Υπάρχουν φυσικά και άλλε πρωτοβουλίε. Φέτο. είχαμε μια σειρά από πλευρές που ασχολούνται και που είπαν ότι θέλουν να κάνουν προτάσεις οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί, ανέφερε την Γαλλική Πρωτοβουλία, πια Βημόν σίγουρα θα την αναφέρει. Ε, θέλω να πω ότι πλήρω τη στηρίζει η Ένωση ευθύ εξ αρχή και ένα από τα επιτεύγματα αυτή τη πρωτοβουλία ήταν ότι βοήθησε. Ούτω ώστε το θέμα αυτό να μείνει στο επίκεντρο τη διεθνού προσοχή, τονίζοντα ακριβώ τη λύση των δύο κρατών. Τώρα, τι κάνει και τι μπορεί να κάνει η Ένωση. Πρέπει να παραμείνουμε εστιασμένοι στις δυνατότητες, στα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να βοηθήσουμε ε, πέραν του κουαρτέτου. Αλλά φυσικά πάντα στο πλευρό των διεθνών εταίρων μας κάνουμε μια σειρά από πράγματα. Κανένα άλλος ε, ε, παράγων που παίζει ρόλο δεν έχει τις δυνατότητες που έχουμε για τη δημιουργία θεσμών, αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια, εκπαίδευση για ε, ε, αποστολές πολιτικού προσωπικού για να εξακολουθεί να παραμένει πράσινη γραμμή, να παραμένει στο χάρτη, να δούμε τι σημαίνει αυτή η γραμμή του 67 ε, εμπλοκή με την ευρύτερη περιοχή, με την πρωτοβουλία την αραβική και για να γίνει πιο λειτουργική, για να χορηγήσουμε κίνητρα και στις δύο πλευρές. Έχουμε αυτή την ειδική προνομιακή εταιρική σχέση που νομίζουμε ότι θα ήταν μια πολύ καλή βάση για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πιο κοντά και με τις δύο πλευρές. Κανένα άλλο δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τα τονίσει αυτά. Πρέπει να τα αξιοποιήσει για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας με τους ε, εταίρους μας. Τώρα περισσότερο παρά ποτέ για τη λύση των δύο κρατών και για να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία. Αυτά όπως είπα, η λέξη είναι να ε, είμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία με όλους, με την εθνική κοινότητα, την νέα Αμερικανική κυβέρνηση και κυρίως ούτω ώστε η διεθνής κοινότητα να παραμείνει ενωμένη γύρω από αυτήν την προσέγγιση των δύο κρατών. Γιατί θεωρώ ότι αυτός θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο πρέσβης Πιέρ θα πάρει τώρα το λόγο. Η Γαλλία προετοιμάζει μία διάσκεψη για τα ζητήματα της περιοχής αυτής. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τις σχέσεις με το κουαρτέτο και τις σχέσεις με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Ίσως αυτό θα μας βοηθούσε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μαζί με τον καθηγητή Βελμέρ και τον κύριο Τζεντιλίνη με καλέσατε σήμερα, με τιμάτε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί ο Φερνάντο είπε ήδη πολλά και δεν θα τα επαναλάβω. Θα ήθελα να προσπαθήσω να εξηγήσω περί τίνος πρόκειται, είναι αυτή η γαλλική πρωτοβουλία και να κάνω και μια έκθεση υπεπραγμένων. Όπως είπε ο Φερνάντο, θα πρέπει να αναζωογονήσουμε, να δώσουμε μια νέα δυναμική στη λύση των δύο κρατών. Νομίζω πως η ειρηνευτική διαδικασία καρκινοβατεί τα τελευταία χρόνια και Εάν θέλει κάποιο κατηγορηματικά να υποστηρίξει αυτή τη λύση, ε, θα πρέπει να αναλογιστεί ότι ήταν ε, κάτι που κανείς δεν αμφισβητούσε πριν από λίγα χρόνια. Κάτι ε, το αυτονόητο. Θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Τονίζω το επίγον του ζητήματος επισημένοντας και άλλους λόγους πέρα από αυτούς που προανέφερε ο Φερνάντο που εξηγούν την κατάσταση επιτόπου. Η νέα ε, Αμερικανική κυβέρνηση και το καθεξής δηλαδή. Ένα στοιχείο που είναι σημαντικό να το θυμόμαστε και σας παραπέμπω και στην πρωινή σας συνεδρίαση για τη Συρία. Σήμερα, όταν ε, κάνετε επαφέ στην περιοχή, είτε μιλάμε για πολιτικούς ηθήνοντες, είτε για την κοινωνία των πολιτών, ε, για ε, προέδρους κομμάτων. Κανείς πλέον δεν μιλά για την ειρηνευτική διαδικασία και την Ισραηλοπαλαιστινιακή σύραξη. Δεν ε, είναι θέμα της επικαιρότητα. Μιλάνε όλοι για τη Συρία, για την Ιεμένη, για τη Λιβύη. η άνοδος των ριζοφαστικών κινημάτων που παρατηρείται σε διάφορες χώρες. Κανείς δεν ασχολείται πλέον με την Μέση Ανατολή και την ενευτική διαδικασία. μέσα αυτή τη κατάσταση αποφασίσαμε να δρομολογήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Είχαμε την αίσθηση πως ε, αφενός είναι επικίνδυνη αυτή η κατάσταση όχι μόνο για τις δύο πλευρές αλλά και για την περιοχή αλλά και για την Ευρώπη και για την ίδια τη διεθνή κοινότητα. Επίσης, η καθεστική τάξη ε, μπορεί να είναι και παραπλανητική. Να μας δώσει την εντύπωση ότι μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως σήμερα και ότι δεν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος αποσταθεροποίησης της περιοχής. Νομίζω όμως η πραγματικότητα μας δείχνει ακριβώς το αντίθετο και ε, αυτός είναι ο στόχος της Γαλλικής Πρωτοβουλίας. Να θυμίσουμε σε όλους πώς. Εάν δεν ε, ξαναπάρουμε αυτό το θέμα στα σοβαρά όπως πριν από λίγα χρόνια, ενδέχεται τους επόμενους μήνες, επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσουμε σοβαρότατα προβλήματα. Αυτή είναι η ουσία λοιπόν της Γαλλικής Πρωτοβουλίας. Έχει ένα διτό στόχο να επαναφέρει αφενός ε, το στόχο, τον, ε, τη λύση των δύο κρατών ε, στο Διεθνές Θεματολόγιο και δεύτερον να το θέσει επιτάπητο στο ζήτημα για να συνεχίσει ο δημόσιος διάλογος και να προκύψουν νέες πρωτοβουλίες και επειδή δεν θέλουμε να σταματήσουμε σε αυτό, να επαναδρομολογήσουμε ε, αυτή την ε, λύση. Όχι να εκκινηθήσουμε μια νέα διαδικασία, διότι υπάρχει ήδη, αλλά να επαναριοθετηθεί ούτω ώστε η λύση αυτή να εξεταστεί στα διάφορα βήματα, στο δίευλο του κουαρτέτου, ε, στις πρωτοβουλίες περιφερειακές από διάφορες χώρες. Η ad hoc Επιτροπή ε, Συνδέσμων που ασχολείται με τα επίγοντα ζητήματα. Να τονίσουμε λοιπόν τη σημασία αυτής της ε, λύσης και να της ε, δώσουμε μια νέα πνοή. Έχουν γίνει και σχετικές δημοσκοπήσεις Ανεξαρτήτως που έγιναν στην Ισραηλινή ή στην Παλαιστινιακή πλευρά, τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Εξακολουθεί να υπάρχει μια ισχυρή πλειοψηφία, δύο τρίτα ε, υπέρ της λύσης, ε, ε, δύο τρίτα των ερωτηθέντων απήντησαν πως η λύση δύο κρατών είναι η μόνη βιώσιμη λύση, όπως έλεγε και ο Φερνάντο. Ταυτόχρονα όμως ισχυρίζεται η ίδια πλειοψηφία ότι δεν είναι ρεαλιστική λύση, δεν είναι δύνατη να υλοποιηθεί και άρα είναι όλο ένα και πιο αφελές να αναφέρει κάποιος ότι είναι μονόδρομος ε, η λύση ε, των δύο κρατών. Δηλαδή οι ελπίδες και η πραγματικότητα χωρίζονται από ένα χάσμα που είναι γόνιμο έδαφος για προβλήματα κρίσης, απόγνωση και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι με την πρωτοβουλία μας ε, θα έπρεπε να υπενθυμίσουμε στη διεθνή κοινότητα, θα πρέπει να συνεχίσει το διάλογο για αυτή τη λύση και να προχωρήσει. Με ποιο τρόπο λειτουργούμε. Η πρωτοβουλία μας διαφοροποιείται σε σχέση με παλαιότερες, γιατί δεν θέλουμε πάση θυσία να ξαναξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ξέρουμε δεν έχει οριμάσει ο χρόνος ακόμη για κάτι τέτοιο. Να ε, τους υποχρεώσουμε τώρα να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Τελικά δεν είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επανεφεύρουμε τον τροχό. Υπάρχουν ήδη ε, διαδικασίες, ε, ε, μηχανισμοί που υπάρχουν και δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε να γίνουν επικαλύψεις. Δεν θέλουμε πάση θυσία να επιβάλλουμε αυτή τη λύση. Η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι επιτόπου για τις σχέσεις των δύο πλευρών και ξέρουμε ότι νέα κυβέρνηση θα αναλάβει σύντομα την εξουσία και θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις. Ε, τι ακριβώς προτίθεται να κάνει. Ενδεχομένως και άλλοι εταίροι να θέλουν να κάνουν κάποια άλλη κίνηση. Δεν θέλουμε επουδενή να επιβάλλουμε μια λύση. Θέλουμε να επιτύχουμε συνένεση, να συμφωνήσουν όλοι για αυτή την ιδέα ότι οφείλουμε και πάλι να ε, δώσουμε τη δέουσα σημασία σε αυτή τη λύση. Και τρίτο στοιχείο δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν. Εξ αρχής είπαμε, όποιος έχει καλές ιδέες, όποιος θέλει να επέμβει, να κάνει κάτι, είναι ευπρόσδεκτος. Επαναδρομολογώντας την, ε, ε, τη, τη, τη λύση αυτή και δίνοντας μια νέα όθηση, στη διαδικασία η Αίγυπτος, η Ρωσία, η απερχόμενη Αμερικανική κυβέρνηση, όπως είπε και ο Φερνάντο, ε, προσπάθησαν να ε, συνεχίσουν τη συζήτηση μετά από αυτή την χρήσιμη ομολογουμένως έκθεση του κουαρτέτου και σήμερα πρωτοβουλία από την Παλαιστινιακή Αρχή για να προχωρήσει με ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τους οικισμούς. Και πάλι, δεν θέλουμε να αποτρέψουμε ε, κανέναν, θέλουμε να συντονιστούμε. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε να, ε, αν υπάρχουν άλλοι εταίροι που θέλουν να ε, συμμετάσχουν. Τι ε, προσδοκούμε, ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα τον Ιούνιο στο Παρίσι, όπως είπατε κι εσείς, Οργανώνουμε αυτή τη διάσκεψη στα πλαίσια τη πρωτοβουλία και μέχρι το τέλος Οργανώσαμε μάλλον συγγνώμη τον Ιούνιο τη διάσκεψη και μέχρι το τέλο του τρέχοντο ε, θέλουμε μία λύση και η νέα διάσκεψη κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει ε, ε, πριν τα Χριστούγεννα. Είναι δύσκολο να βρούμε μία ημερομηνία, πάντως σε αυτή τη διάσκεψη ε, τρεις στόχους θα έχουμε. Πρώτον, Ισχυρή πολιτική δέσμευση από όλους τους συμμετέχοντες. Ισχυρή πολιτική δέσμευση για την λύση των δύο κρατών και για τις αρχές στις οποίες εδραιώνεται αυτή η λύση και τις κατευθυντήριες γραμμές, τους όρους που έχουν εγκριθεί επανειλημμένα από το 67 είτε μιλάμε για το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ε, τον δικό χάρτη του κουαρτέτου, άλλα έγγραφα και ε, η πρόσκληση από τον James Baker προς την ε, διάσκεψη της Μαδρίτης, πολύ σημαντικό έγγραφο, πολύ σημαντικό διάβημα και υπάρχει μια σειρά από τέτοια έγγραφα. Λοιπόν, αυτή την διάσκεψη θα τη χρησιμοποιήσουμε ούτως ώστε να ρίξουμε τα θεμέλια για την αναζωογόνηση αυτής της λύσης. API επίσης, ε, αραβική πρωτοβουλία, ειρηνευτική πρωτοβουλία, αναφέρθηκε και ο Φερνάντος αυτή, έχει ε, αποτελματωθεί αυτή τη στιγμή και θέλουμε και πάλι να δώσουμε μια νέα πνοή σε αυτήν την αραβική πρωτοβουλία, διότι ε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ε, για συνενέσεις, ε, για αμοιβαία κατανόηση για τους, τους εταίρους της περιοχής αυτής. Θα θέλουμε να προσπαθήσουμε να πιέσουμε χωρίς όμως να ζητήσουμε νέες παραχωρήσεις από οποιαδήποτε πλευρά, διότι δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Αυτό που θέλουμε είναι θα, να συνεχίσει η Ραβική Πρωτοβουλία, διότι υπάρχει εδώ και χρόνια, χωρίς όμως να έχουν συμβεί πολλά πράγματα, χωρίς να έχει αυτά αποτελέσματα. Επίσης, να έχουμε τις ε, προσφορότερες προϋποθέσεις μέσω συγκεκριμένων ρεαλιστικών προτάσεων επιτάπητος, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα επιτρέψει σε αυτήν την λύση των δύο κρατών να αποκτήσει μια νέα ζωή. Η οικονομική ανάπτυξη, πως οι εταίροι ε, θα αντιληφθούν ότι η διεθνή κοινότητα είναι σε εγρήγορση, προτίθεται να βοηθήσει τους ώστε να ε, δημιουργήσει το ε, προσφορότερο οικονομικό περιβάλλον για να προχωρήσει και η πρωτοβουλία για τη λύση των δύο κρατών. Μιλώντας για την οικονομική κατάσταση στα Παλαιστινιακά εδάφη και εκεί καρκινοβατούμε, βλέπουμε για την ανάπτυξη παραδείγματος χάρη για το δημόσιο έλλειμμα, για την ανεργία κτλ. Ε, ε, μεγέθη που ε, δυστυχώς φθήνουν. Και εκεί θα πρέπει να δράσουμε η Παλαιστινιακή Αρχή επίσης θα πρέπει να εδραιώσει την ικανότητα διακυβέρνησης που έχει. Υπάρχει διεθνή αρρωγή, αλλά με ποιο τρόπο μπορεί να είναι καλύτερα στοχοθετημένη, καλύτερα συντονισμένη για να επικουρεί την Παλαιστινιακή πλευρά. Ε, είμαστε στενές επαφές και συνεργασία με τους Παλαιστινίους, ούτως ώστε να νιώθουν ότι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της νέας κατάστασης. Και ξαναλέω ότι πρέπει να ζωγονηθεί ο δημόσιος διάλογος και στις δύο πλευρές για τους λόγους που προανέφερα. Ε, οι οργανώσεις τη κοινωνίας των πολιτών έχουν χάσει την πίστη, την εμπιστοσύνη τους στη διαδικασία και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, να παροτρινθούν, να μετάσχουν ε, ούτω ώστε να ε, αρχίσει ο δημόσιος διάλογος και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη. Και το τρίτος στόχος που επιδιώκουμε από αυτή τη διάσκεψη είναι να γίνει ένα σωστό follow Ε, και αναμένεται να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες ε, είναι ένα δίευλη επικοινωνία ε, το κουαρτέτο, το Σύμβουλο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η ρωσική πλευρά, η νέα Αμερικανική κυβέρνηση να συμμετάσχουν στη διαδικασία, να, στο πλευρό μας, να, οθεί, να δώσουμε μια νέα όθηση σε αυτή τη διαδικασία για να επανεγγραφεί ε, στο Διεθνές Θεματολόγιο αυτή η λύση. Αν δείτε επιτόπου ποιες συζητήσεις γίνονται, θα ανακαλύψετε ότι σίγουρα ε, τη σήμερα ημέρα είναι ε, η μεγαλύτερη πρόκληση στην οποία πρέπει να αντεπεξέλθουμε. Αν επανδρομολογήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, τότε θα υπάρχουν ελπίδες ότι η ειρηνευτική διαδικασία θα αναζωογονηθεί και θα ε, συνεχίσει με ανανεωμένη ενέργεια. Θα σταματήσω εδώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο καθηγητής Μπεν τώρα. Έχετε δει πάρα πολλέ ε, ήττε σε ό,τι αφορά τι ελπίδε Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Με τιμά να είμαι εδώ μαζί με τον ε, κύριο Βημόν και τον κύριο Τζεντιλίνη. Είχα την ικανοποίηση να συναντηθώ με αυτούς τους κυρίους πάνω από δύο φορές και εκτιμώ όλα όσα υπόθηκαν και συμφωνώ με πολλά από τα σημεία που τέθηκαν σήμερα αλλά και στο παρελθόν αλλά θα ήθελα να κάνω ένα βήμα προς τα πίσω και να επανέλθω στην αρχή της ε, λύσεις των δύο κρατών. Γιατί μιλάμε ότι αυτή είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή. Αυτό έρχεται από την πολύ βασική αρχή, την συνύπαρξη. Δηλαδή οι Ισραηλοί και οι Παλαιστίνοι συνυπάρχουν, είτε τους αρέσει είτε όχι. Η συνύπαρξη είναι αναπόφευκτη και ε, αυτό υπό τις καλύτερες ή χειρότερες συνθήκες. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει λύση των δύο κρατών, δεν θα είναι δυνατή η συνύπαρξη και δεν θα μπορούν να διατηρούν επαόριστον Ισραηλινή την κατοχή και αυτό γιατί ακριβώς πρέπει να υπάρχουν και οι δύο πλευρές και δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Αλλά να σας εξηγήσω τις δυσκολίες. Θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα στους αυτούς μας γιατί μετά από 50 χρόνια, από το 1967, 70 χρόνια μάλλον, γιατί οι λαοί δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Αυτή είναι η βασική αρχή που χρήζει απάντησης και θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση σε δύο στάδια, τι έχουμε, ποιες είναι οι άμεσες συνθήκες στη Μέση Ανατολή. Εγώ πιστεύω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων σήμερα, δηλαδή να ξανακαθίσουν στο τραπέζι, θα αποτύχουν. Θα αποτύχουν γιατί θα πρέπει να δούμε εντάχει την κατάσταση και στο Ισραήλ και στην περιοχή. Καταρχήν η Ισραηλινή κυβέρνηση σήμερα δεν είναι δεσμευμένη για αυτή τη λύση των δύο κρατών. Πρέπει να δούμε, αρκεί να δούμε τη σύνθεση της κυβέρνησης στο Ισραήλ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που καλούν να υπάρξει ένα τέλος στην ιδέα των, ε, της λύσης των δύο κρατών ε, και μάλιστα ζητάνε την προσάρτηση της δυτικής όχθης κυρίως της περιοχής ΣΥ. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει δέσμευση εντός αυτής της ε, κυβέρνησης στο Ισραήλ. Επίσης πρέπει να δούμε την Ισραηλινή αντιπολίτευση. Σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματική αντιπολίτευση στο Ισραήλ που να μπορεί να αντιμετωπίσει σήμερα την κυβέρνηση μετά το 2019 ήταν λίγη θητεία της σημερινής κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν, καθώς ε, οι άνθρωποι μετακινούνται περισσότερο στο Ισραήλ προς τα δεξιά και την κεντροδεξιά, έτσι λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το εμπόδιο. Το τρίτο που θέλω να αναφέρω είναι το αραβικό κράτος. Σήμερα τα αραβικά κράτη. Τα αραβικά κράτη θα ήθελαν να δουν να υπάρχει ένα τέλος της σύραξη, αλλά ανησυχούν με τα δικά τους θέματα εσωτερικής ασφάλειας βλέπουμε ότι τα κράτη του κόλπου, τα αραβικά κράτη είναι σε συχνέ επαφέ με το κράτος του Ισραήλ γιατί από τη δική του σκοπιά το Ισραήλ ουσιαστικά αποτελεί το προμέτωπο για την ε, άμυνα απέναντι στο Ιράν και δεν χρειάζεται να πιέσουν γιατί σε ό,τι αφορά αυτούς ε, μπορεί το ζήτημα το να μπει σε δεύτερο επίπεδο, είναι χαμηλή προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν δεν είναι έτοιμοι απαραίτητο να καθίσουν και να δώσουν αυτή την όθηση στη διαδικασία. Κατόπιν πρέπει να δούμε την Παλαιστινιακή Αρχή και πρέπει να σας προτείνω δυστυχώς ότι σήμερα δεν υπάρχει ηγεσία στην Παλαιστινιακή Αρχή που μπορεί να φέρει τα απαραίτητα αποτελέσματα και να κάνει τις υποχωρήσεις για την επίτευξη της συμφωνίας. Η Παλαιστίνη είναι κατακαιρματισμένη, όσο και το Ισραήλ υπάρχει Χαμάς, η Παλαιστινική Αρχή δεν ε, βλέπουν ε, πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουν στο ίδιο επίπεδο και θα προσεγγίσουν τη σύραξη. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε σημαντική κίνηση από την πλευρά της Παλαιστινιακής Αρχής. Και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω, που θα έπρεπε να ήταν το πρώτο, είναι η θέση της νέας κυβέρνησης. Τραμπ όταν θα αναλάβει ο Τραμπ τις επόμενες εβδομάδες ε, δεν έχει συγκεκριμένη θέση για το ζήτημα. Δεν ξέρουμε ακριβώς ε, ποια θέση θα λάβει η νέα κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στο Πανιστιακό. Όμως ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα εμπλακεί σε κάποια διαδικασία αν δεν υπάρχει καλή πιθανότητα επιτυχίας θα είναι σαφής, θα αξιολογήσει τη σύραξη πριν να αναλάβει δεσμεύσεις ε, για να ξεκινήσει διαδικασία. Όμως, εν τω μεταξύ, θα συνεχίσει να ακολουθεί τα χνάρια των προκατόχων του, δηλαδή σίγουρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Ισραήλ. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να αναζωογονήσουμε αυτό το ζήτημα, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει οπωσδήποτε η στήριξη των Αμερικανών, γιατί χωρίς την αμερικανική στήριξη και την άμεση συμμετοχή των Αμερικανών, η διαδικασία δεν θα κινηθεί προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Όμως το τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι ίσως το πιο σημαντικό και έχει συζητηθεί πολύ λίγο στο παρελθόν και αυτό είναι η ψυχολογική διάσταση του Ισραηλοπαλαιστινιακού. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πέραν των όσων πιστεύουμε και πέρα από τα πρακτικά βήματα που θα πρέπει να γίνει προκειμένου να κινηθεί προς τα μπρος η διαδικασία, υπάρχουν ψυχολογικά εμπόδια που καθιστούν αδύνατο και για τις δύο πλευρές να κάνουν τις απαραίτητες παραχωρήσεις, ε, παρόλο που ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν αυτές τις υποχωρήσεις. Πώς ε, θα αλλάξει σε την ιστορική αφήγηση, πώς ε, θα αντιμετωπίσει το θρησκευτικό ζήτημα Πώς ε, θα αντιμετωπίσει την ιδεολογική εφήγηση. Οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές έχουν ε, ουσιαστικά υιοθετήσει ένα διαφορετικό δόγμα και δεν είναι σε θέση να κάνουν τις απαραίτητες υποχωρήσεις γιατί πάντοτε τους έλεγαν ότι δεν θα συμβεί. Λένε Ισραηλινοί, η Ιερουσαλήμ θα μείνει αιωνίω η πρωτεύουσα του Κράτου τη Ισραήλ. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μέρο του Παλαιστινιακού κράτου. Και οι Παλαιστινοί θα συνεχίσουν να επιμένουν ε, στο δικαίωμα τη επιστροφή. Έχουμε ζητήματα εδώ που ξέρουμε ότι πρέπει να συμβούν, ε, αλλά ε, το έχει υιοθετηθεί ένα συγκεκριμένο δόγμα από το ΛΟΚ. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν αυτή η δημόσια φυγή, προκειμένου να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα σημειωθεί καμία πρόοδος ανεξάρτητα από τις προσπάθειές μας. Επομένως, πρέπει να σας προτείνω ότι πριν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να σκεφτούμε σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της συμφιλίωσης. Για μένα αυτό είναι προϋπόθεση για την επιτυχία στο μέλλον. Η διαδικασία της συμφιλίωσης απαντά σε τρεις βασικές ερωτήσεις. Καταρχήν, σε τρία ζητήματα. οικοδόμηση εμπιστοσύνη καταρχήν. Σήμερα είναι μηδενική εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα από λαό σε λαό και άλλα μέτρα για να είμαστε σίγουροι ότι αρχίσουμε να μετριάζουμε αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνη. Το δεύτερο είναι το αμοιβαίο αίσθημα ανασφάλεια σε οποιαδήποτε διαδικασία συμφιλίωσης θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πώ θα νιώσουν πιο ασφαλείς οι Ισραηλινοί και πώ θα νιώσουν και πιο ασφαλεί οι Παλαιστίνοι. Δηλαδή αυτή η έννοια τη ανασφάλεια και από τι δύο πλευρέ προκαλεί πολλού δισταγμού για το πώ θα προχωρήσουν. Και το τρίτο σημείο που θα πρέπει να μετριαστεί, να βληθεί, είναι οι ψευδεστήσει που κάποιοι Ισραηλοί και Παλαιστινοί συνεχίζουν να θερέφουν ότι μπορούν να έχουν τα πάντα. Έχουμε από τη μία τη Χαμάς ε, και τους ε, πολύ δεξιούς Ισραηλινούς ε, που λένε είναι δική μας γη. Αυτοί δεν είμαστε έτοιμοι να τη διαιρέσουμε ούτε να εγκαταλείψουμε οποιοδήποτε μέρο της. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε αυτές τις ψευδεθήσεις, να διαλύσουμε αυτές τις ψευδεθήσεις και από τις δύο πλευρές έτσι ώστε να καταλάβουν ότι είναι αναπόφευκτη συνύπαρξη και κανείς δεν μπορεί να τα έχει όλα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια διαδικασία συμφιλίωσης και η διαδικασία της συμφιλίωσης σημαίνει τρία πράγματα δηλαδή να έχουμε δράσεις από λαό σε λαό. Εγώ δεν έχω χρόνο τώρα να αναφερθώ λεπτομερώς, αλλά ευχαρίστω να απαντήσω στο θέμα αυτό. Το δεύτερο είναι διαδικασία, για τη διαδικασία της φελίωσης είναι ότι οι σημερινές κυβερνήσεις και οι δύο μπορούν να κάνουν περαιτέρω βήματα για να αμβλύνουν την ένταση και την πίεση. Πολλά παραδείγματα μπορούν να δοθούν, χάρη, και για τις δύο πλευρές, χωρίς να γίνει, παραδείγματος χάρη, κάποια σημαντική παραχωρήση που δεν είναι έτοιμη να τη κάνουν. Και η τρίτη οδός πρέπει να βασίζεται στο πιο πολιτικό πλαίσιο θα πρέπει να προωθηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συμφιλίωσης που μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον δύο χρόνια. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η ειρηνευτική πρωτοβουλία μας. Αυτό πρέπει να είναι το γενικό πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνική πρωτοβουλία, γιατί οποιαδήποτε πρωτοβουλία δεν έχει πλήρη εκπροσώπηση των αραβικών κρατών, δεν θα πετύχει. Πολλοί από εμά ε, ξεκολουθούν να πιστεύουν ότι το κορτέτο θα δώσει ένα μέρο τη απάντηση. Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι αν θέλουμε να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά και θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία και στο πλαίσιο αυτό σίγουρα η Γαλλική Πρωτοβουλία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Για να πάω τώρα στη Γαλλική Πρωτοβουλία και να πω με σαφήνεια προσωπικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, θα πρέπει να επιδιωχθεί και να λάβει χώρα. Το ερώτημα σήμερα είναι πότε και ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτής της διάσκεψης. Αναμφίβολα, με τις καλύτερες προθέσεις, ο κύριος Βημών θα ήθελε να λάβει χώρα αυτό τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες. Κατά την άποψή μου, το να ε, πιέσουμε για να γίνει μια τέτοια διάσκεψη πριν τα Χριστούγεννα, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι σκέφτεται η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση Τραμπ, θα είναι αντιπαραγωγικό. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούμε για κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύω κάθεται ότι η γαλλική πρωτοβουλία από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αποτύχει. Θα πρέπει να αποτρέψουμε την αποτυχία με κάθε κόστος. Γιατί εάν αποτύχετε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθουμε και να προσπαθήσουμε να ξαναδώσουμε νέα πνοή στη διαδικασία ενώ θα έχουμε μία αποτυχία που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί καταρχήν. Το δεύτερο είναι τι θα πρέπει να είναι στην ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να επικεντρωθεί στην διαδικασία. Τι θα κάνουμε τα επόμενα δύο χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα μπορέσει να επικεντρωθεί στην αστροπινιστική σύραξη για κάποιο καιρό. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πάρα πολλά άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσει, πιο ή πιο επίγοντα, κατά την απόψή του, και εφόσον ε, δεν ε, είναι επίγουσα η σύραξη αυτή, θα τεθεί κατά μέρου. Και αυτό δίνει μια ευκαιρία για την Γαλλική Πρωτοβουλία να εκμεταλλευτεί την περίοδο αυτή για τους επόμενους 18 μήνες με δύο χρόνια για να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, να προετοιμάσει το έδαφος για μια επακόλουθη σειρά διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μερών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γαλλική Πρωτοβουλία είναι κρίσιμη σημασίας για να αναλάβουν αυτό το ρόλο και να προετοιμάσουν το έδαφος για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η Γαλλική Πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντική, όμως κάποια βήματα θα πρέπει να γίνουν μαζί με την προετοιμασία του εδάφους. Θέλω να φέρω ένα-δυο παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ θα εναγκαλύψει την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία. Αυτή είναι μια σημαντική κίνηση προς τον μπρος. Ήδη ο Νετανιάχου έχει πει ότι του αρέσουν κάποια στοιχεία αυτή τη πρωτοβουλία. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειε να πείσουμε τη Χαμά να εναγκαλίσει την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία και μπορούμε να στραφούμε στο κατά στην Τουρκία και άλλου που έχουν πολύ καλέ σχέσει με τη Χαμά για να τι εξηγήσουν γιατί είναι απαραίτητο να, κινηθούν προ αυτή την κατεύθυνση, γιατί ε, δεν πρόκειται να συμβούν αυτά που ονειρεύονται. Πρέπει να γίνει προσπάθεια για να μετριάσουμε και αυτό το πρόβλημα. Γιατί όσο η Χαμάς και άλλες εξτρεμιστικές ομάδες συνεχίζουν να καλούν για την καταστροφή του Ισραήλ, τότε ουσιαστικά εξυπηρετούν ε, την Ισραηλινή κεντροδεξιά και για πολύ καλό λόγο θα σας πούν γιατί να κάτσουμε να διαπραγματευτούμε για να κάνουμε σοβαρές υποχωρήσεις ενώ θέλουν να μας καταστρέψουν. Έτσι λοιπόν, ε, στο πολιτικό επίπεδο πρέπει να γίνει πολλή δουλειά από τους Γάλλους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος και πάλι σε επίπεδο λαών, λαό σε λαό, κυβέρνηση με κυβέρνηση και να υπάρχει και ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και ιδίως από τα αραβικά κράτη. Και αν μπορούμε ε, σε αυτό να βάλουμε και το Ισραήλ και τη Χαμάς να συμμετέχουν, και θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία που και τα δύο μέρη θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από σήμερα μέχρι τα επόμενα δύο χρόνια δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά εγώ μπορώ να σα πω κατηγορηματικά κατά την άποψή μου ότι η σημερινή ηγεσία στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη δεν είναι σε θέση, ούτε θα είναι σε θέση να παράξουν αποτελέσματα, να κάνουν κάποια σημαντική υποχώρηση για να προχωρήσει η διαδικασία. Και γι' αυτό το λόγο τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε ως όχημα τη γαλλική πρωτοβουλία. Ένα επιτυχές όχημα για να προετοιμάσουμε το έδαφος προς αυτό το σκοπό. Και αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία δεδομένη τη κατάσταση στι Ηνωμένε Πολιτείε και τη πραγματικότητα στην ίδια τη Μέση Ανατολή, δεδομένου του γεγονότο ότι καμία πλευρά δεν είναι έτοιμη να κάνει τι απαραίτητε υποχωρήσει. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Γάλλοι μπορούν να παίξουν ένα σημαντικότατο ρόλο για να δώσουν όθηση στη διαδικασία και όταν έρθει ο καιρός, 18 μήνες, 2 χρόνια, θα δούμε να υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή από τις δύο πλευρές να ακούσουν. Σε σχέση με το γιατί η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη πρακτική λύση που τελικά θα δώσει στο Ισραήλ είναι έσχατη ασφάλεια και θα καλύψει και τις προσδοκίες των Παλαιστινίων καθώς χρειάζονται ένα ελεύθερο δημοκρατικό κράτος για να ζουν ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ. Αυτό δεν είναι ένα ψευδές όνειρο, μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για να κινήσουμε τη διαδικασία και όχι τώρα να έχουμε ψευδεστήσεις και να λέμε στους ανθρώπους αυτούς ελάτε να κάτσετε να ξεκινήσετε τις διαπραγματεύσεις και είδαμε που απέτυχε η κυβέρνηση Ομπάμα. Γιατί κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, Ισραηλοί, Παλαιστίνοι, Ηνωμένε Πολιτείε δεν σκέφτηκαν προσεκτικά τι χρειάζεται να γίνει για να αλλάξει την αντίληψη, την οτροπία της κοινή γνώμης και να την προετοιμάσει να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δουν ο ένας τον άλλον ως εταίρο για την ειρήνη, ως γείτονες που μπορούν να ζήσουν ειρηνικά με ασφάλεια. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και πιστεύω ότι είναι δυνατόν να συμβεί εφόσον έχουμε ένα πολύ προσεκτικό πλαίσιο προς αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βλέπω τις αντιφάσεις ε, στα επιχειρήματα δύο εκ των ομιλητών. Ο πρέσβης Τζεντιλίνη και ο καθηγητής Μπεν Μέιρ. Διότι ο κύριος Τζεντιλίνη τόνισε τη σημασία της αμερικανικής στήριξης προς την ερνηφτική διαδικασία. Ενώ ο καθηγητής ε, τόνισε ότι προς το παρόν, λόγω της αλλαγής πολιτικής και κυβέρνησης, είναι απούσες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το θεωρεί μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα πιο αποφασιστικό ρόλο, να έχει μεγαλύτερη επιρροή. Εγώ, με βάση όλα όσα γνωρίζουμε, έχω τις αμφιβολίες μου. Και θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο το εξής. Ε, πώς ε, προβλέπετε ότι θα ε, αναπτύξει την πολιτική του ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή και τι θα γίνει με τη λύση των δύο κρατών. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ο κύριος Παγνιού. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους κυρίους ε, Ζωντιλίνη, Βημό και Μελμέρ για τις ε, παρουσιάσεις σας. Νομίζω ότι είναι σωστή στιγμή. Λίγες εβδομάδε πριν από τη Νέα Γαλλική Πρωτοβουλία, όπως είπε ο Πιέρ και λίγες εβδομάδε μετά την εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ και τις μεγάλες αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλεί όπως ε, υπενθύμησε ο κύριος Μπένμερ, ευχαριστώ για την απάντηση του Πρόεδρου Μπρόκ που συμφώνησε μετά από πρότασή μου να οργανώσουμε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων ε, πολύ σύντομα. Ο επόμενος χρόνος είναι ένας χρόνος πολύ σημαντικός που θα έχει διάφορες συμβολικές ημερομηνίες. 100 χρόνια από την διακήρυξη Μπάλφουρ, 70 χρόνια από το σχέδιο ε, δικοτόμης ε, Παλαιστίνης και 50 χρόνια από το ψήφισμα 142. Το 2017 είναι συμβολικό λοιπόν. Περισσότερο παραποτέ μας καλεί να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις, όπως ε, τις παρουσιάσατε. Αλλά πρέπει να σημειώσω ότι η εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ αλλάζει την τράπουλα. Ε, μπορεί όμως να αποτελεί ευκαιρία για την Ευρώπη, εφόσον είναι σαφές ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, δεν είναι διατεθειμένες να ασχοληθούν με την επίλυση αυτού του προβλήματος, αυτής της σύραξη. Άρα η δική μας ευθύνη είναι μεγαλύτερη παραποτέ. Και αυτό υπόθηκε σε σχέση με τη Γαλλική Πρωτοβουλία. Τέσσερις ερωτήσεις κύριοι. Πρώτον, το θέμα σήμερα, είτε είναι κανείς Παλαιστίνιος είτε Ισραηλινός, είναι οι ηγεσίε. Ούτε ο Νετανιάχου, ούτε ο Μαχμούντα Μπάς έχουν την ε, δυνατότητα να επιβάλλουν μια λύση. Οποιαδήποτε ειρηνευτική λύση θα οδηγούσε στην κατάρρευση των κυβερνήσεων που θα το υπέγραφαν. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αρκεί απλώ να καθίσουν στην τράπεζα να το πραγματεύσουν. Το υπενθύμησε ο Αλόν Μπερμέρ. Πώ προβλέπετε λοιπόν μια πρωτοβουλία, όπω η Γαλλική Πρωτοβουλία θα μπορούσε να βοηθήσει με τη στήριξη τη Ένωση. Πώ θα μπορούσε δηλαδή να δημιουργήσει τι συνθήκε για να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει κατάλληλη πολιτική ηγεσία για να υπάρξει μια νέα όθηση σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία που όλοι θέλουμε. Δεύτερον, η λύση των δύο κρατών ε, είναι φιλόδοξος ε, πολιτικός στόχος επειδή ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση, η επέκταση των οικισμών μειώνει όλο και περισσότερο τη δυνατότητα επιβίωσης ενός παλαισθηνιακού κράτους. Η τελευταία έκθεση του κουαρτέτου ήταν σαφής. Πώς θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αλλάξει την κατάσταση, να σταματήσει τους επικισμούς. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να υπάρξει μια λύση δύο κρατών. Τι κάνουμε για τη σήμανση των προϊόντων από τους επικισμούς. Ιδιαίτερα μετά τις κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο. Τρίτη ερώτηση. Όσον αφορά αυτή τη διάσκεψη που θα οργανώσει η Γαλλία το θέμα της σα διάταξη οπωσδήποτε θα είναι κρίσιμο. Ανάλογα με το τι ακριβώ θα συζητηθεί θα αποφασίσει αν θα έρθει το Ισραήλ. Γιατί ξέρουμε ότι ο κύριο Νετανιαχού ήδη πιέζεται από άλλα μέλη τη κυβέρνηση του να μην συμμετάσχει. Κύριε Βημόν, μπορείτε να μα πείτε περισσότερα από αυτού. Πώ μπορούμε να επιτύχουμε μια συμφωνία για να ξέρουμε αν θα έρθει ή όχι ο κύριος Νετανιάχου. Και επίση είναι σαφέ η επανεκκίνηση της ε, ειρηνευτική διαδικασίας περνάει από την Αραβική Πρωτοβουλία. Αυτή θέτει ένα αρκετά λογικό πλαίσιο για να επανέλθουν όλοι στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Πρέπει λοιπόν ε, αυτή η πρωτοβουλία που είναι από το 2002 να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκε. Γιατί θεωρώ ότι ορισμένε Αραβικέ χώρε διστάζουν να την προσαρμόσουν στι σημερινέ συνθήκε. Έχουμε λοιπόν επαρκή. Ε, δυνατότητες για να υπάρξει μια αποδεκτή νέα αραβική πρωτοβουλία, αποδεκτή και από το Ισραήλ και από τις αραβικές χώρες. Γιατί αν δεν πετύχουμε όλα αυτά, τότε θα έχουμε το σύνολο των αραβικών χωρών και το Ισραήλ που θα συμφωνούν επί ενός κοινού πλαισίου δυστυχών. Άρα θα μειωθεί η δυνατότητα παρενόχλησης από τις πιο ακραίες πλευρές Ισραηλινές ή Παλαιστινιακές όπως είπε και ο κ. Μπενέρ. Και τώρα ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα επιτύχουμε την ειρήνη. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Διότι η κατάσταση μόνιμης σύραξης ε, είναι ανυπόφορη για πολλούς. Το Ισραήλ δημιουργήθηκε ούτως ώστε να εγγυηθεί την ειρήνη για τον Ισραηλινό λαό. Η σημερινή κατάσταση λοιπόν είναι αφόρητη για τους ε, Εβραίους στο Ισραήλ αλλά και για, τους, ε, για την ε, μειονότητα μουσουλμάνων Αράβων. Η προοπτική λύσης δύο κρατών είναι η μόνη που μπορεί να προωθηθεί. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και για την χριστιανική μειονότητα στον αραβικό κόσμο. Μόνο εάν προωθήσουμε την ειρήνη μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ειρήνη. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, σήμερα έχουμε επιλέξει, κατά τη γνώμη μου, την ε, χείριστη οδό. Έχουμε διεθνοποιήσει το θέμα της ειρήνης ε, στους Αγίους Τόπους. Προσπαθούμε να πείσουμε και τις δύο πλευρές, και την Αραβική και την, ε, και την ότι όλα είναι καλά και ότι οι εταίροι τους είναι αξιόπιστοι. Κάποιοι Ισραηλινοί υπουργοί εκφράζονται υπέρ της λύσης δύο κρατών, αλλά στη Γάζα ε, την εξουσία την έχει στα χέρια της η Χαμάς. Έχει γίνει ένα εντελώς πολιτικοποιημένο έδαφος η λωρίδα της Γάζας και όπως ξέρετε δεν υπάρχει ε, κανένα σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ούτω ή άλλω επικίνδυνη αυτή η κυβέρνηση η Χαμά και για τι μειονότητε στη δική τη την ε, περιοχή. Αλλά δεν τα αναφέρουμε όλα αυτά, δεν τα συζητάμε. Α υποθέσουμε ότι δημιουργείται Παλαιστινιακό κράτο. Αυτό το κράτο από την ώρα μηδέν τη ίδρυσή του θα είναι αποτυχημένο κράτο. Κράτο που θα έχει καταρρεύσει. Ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι ε, δεν συμφωνώ. Ε, δεν συμφωνούν μαζί μου, συγγνώμη. Αλλά το βασικό είναι ότι πρέπει να καταλάβουν και οι δύο πλευρές τι πραγματικά χρειάζονται. Χρειάζονται πραγματικά δημοκρατικά καθεστώτα. Πρέπει να έχουν αντιπροσωπευτική δημοκρατία που να αναγνωρίζεται και να έχει αξιοπιστία έναντι της κοινωνίας. Πρέπει να υπάρχει κοινωνική ειρήνη. Επαραλαμβάνω. Η διεθνοποίηση του θέματος αυτού δεν είναι η σωστή οδός, διότι δημιουργεί ψευδεστήσεις. Έχει κανείς την εντύπωση δηλαδή, αν μελετήσει επιφανειακά το θέμα, ότι οι δύο πλευρές έχουν αξιόπιστους συνομιλητές που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη. Η ειρήνη στους Αγίους Τόπους μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν υπάρξει περισσότερη κατανόηση, αλληλοκατανόηση των πλευρών. Φυσικά η διεθνή κοινότητα είναι επίσηματική, αλλά δεν θα πρέπει να ασκεί ε, υπερβολικές πιέσεις επί των ε, δύο πλευρών επιτόπου, γιατί έτσι απομακρύνουμε την προοπτική ειρήνης. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάουτμαντς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους, αλλά Δυστυχώς δεν είμαι ικανοποιημένη και δεν νομίζω ότι θα βρούμε λύσεις για το μέλλον με τη σημερινή συζήτηση. Έχω συγκεκριμένα ερωτήματα. Με την κυρία Μογκερίνη συζητήσαμε ακριβώς αυτό το θέμα στο Στρασβούργο και έθεσα κάποια ερωτήματα και θα ήθελα να σας τα θέσω και σας πρώτο. Κανείς από εσά ε, δεν μίλησε για τα projects που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που καταστρέφονται αυτή τη στιγμή. Εγώ έμαθα ότι αυτός που καταστρέφει κάτι πρέπει να φέρει και το κόστος. Δεν πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε αποζημίωση για τα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να ε, γίνει μια επανόρθωση των ζημιών. Θέλω την απόψή σας γι' αυτό. Δεύτερον, υπάρχει μια σειρά από ειρηνευτικές πρωτοβουλίες όμως ε, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος και το τονίσατε κι εσείς. Ούτε καν συντονισμό δεν υπάρχει ανάμεσα στι διάφορε πρωτοβουλίε. Μήπω ε, σε αυτό έγκυται ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Μογκερίνη, για να συνδυαστούν αυτέ οι πρωτοβουλίε, ε, ούτω ώστε να προκύψει ένα αυθεντικό σχέδιο δράση συγκεκριμένο με προθεσμίε. Γιατί αλλιώ θα παραταθεί αέναο ε, η σύγκρουση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Thank you, Mrs. Chairwoman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τίνω να πιστέψω ότι ακαδημαϊκές συζητήσεις κάνουμε εδώ, γιατί δεν υπάρχει ε, μόχλευση, δυνατότητα άσκησης πίεσης για να υπάρξει πρόοδος. Ε, το ίδιο θα έλεγα και για τους panelists. Συγχαίρω τον εκπρόσωπο της Γαλλίας, ε, τον για την ε, πρωτοβουλία, όμως συμφωνώ με τον καθηγητή. Είναι προώρη αυτή η κίνηση. Ίσως θα έπρεπε να αναβληθεί τουλάχιστον. Υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε ευθαρσός να πει ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί καμία λύση. κυρίως τώρα με την εκλογή του νέου Πρόεδρου, τον είπα, θεωρούν ότι νομιμοποιούνται να συνεχίζουν ε, στον ίδιο δρόμο, να κατεδαφίζουν σπίτια. Χιλιάδες Παλαιστινίους να τους διώχνουν από τα σπίτια τους. Πάνω από 1.500, πρόσφατα μόνο. Να χτίζουν νέους οικισμούς. στις ζώνες όπου ζούσαν οι Παλαιστίνοι μέχρι τούδε. Ακόμη και κτίρια κατεδαφίζουν που ε, οικοδομούνται με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, στη θέση τους ε, ορθώνονται οικισμοί για τους επίκους. Ρωτώ λοιπόν, Κανείς δεν θα βρεθεί να πει πως οι δυνάμεις που υποστηρίζουν το Ισραήλ και τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει αυτή την κατεύθυνση και το είπε και ο καθηγητής ότι ίσως η Τουρκία έχει, μπορεί να ασκήσει πίεση ε, στη Χαμάς ε, να τους υπαγορεύσει τι θα κάνουν. Μα δεν βλέπετε ότι θα γίνει κράτος της Χαμάς η Τουρκία σύντομα. Πώς μπορείτε να περιμένετε ότι θα δώσουν ε, ε τις σωστές συμβουλές. Και επειδή είπατε ότι ε, απεργάζεται την καταστροφή του Ισραήλ η Χαμάς, τότε δεν μπορεί να προκύψει λύση. Όμως ακούστε με, Συμφωνώ ότι αυτά λέει Χαμάς, αλλά αυτοί που το πράττουν είναι οι Ισραηλινοί κατά των Παλαιστινίων. Αυτοί δρούν συγκεκριμένα για την καταστροφή των Παλαιστινίων. Και να προσθέσω επίσης ότι η ΕΣΑΗ λύση δεν θα προκύψει. Θυμηθείτε όμως ότι στις επιθέσεις των Ζελινών κατά τις ε, Λωρίδας Γαζα δύο χρόνια πριν, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 300 άνθρωποι, πάνω από 3.000, για δύο μήνες ε, κρατούνταν και να μην ξεχνούμε ότι γεννήθηκαν αντίστοιχα, αντίστοιχα, γεννήθηκε αντίστοιχος αριθμός Παλαιστινίων κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ευχαριστούμε κύριο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτές τις εξηγήσει ενδιαφέρουσες μένα αλλά απογοητευτικές δε, κυρίως σε σχέση με τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα, εντάξει υπάρχουν γεωπολιτικές αναλύσεις, ε, μια σειρά λόγων ε, που εξηγήσατε με έξοχο νεοτετρόπο για την πραγματικότητα που επικρατεί επί τόπου. Εγώ όμως θέλω να επανέλθω στην ικανότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είμαστε στο Κοινοβούλιο, στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει συγκεκριμένα σε διάφορους τομείς. Από τις εξηγήσει που μας δώσατε, ε, αντιλαμβάνομαι ότι ε, είναι επιτακτική ανάγκη να αναβαθμιστεί η ειρηνευτική διαδικασία. Ίσως ε, απατώμε και διορθώστε με, αλλά έχω την εντύπωση πως ε, ένας από τους εταίρους Ένωσης, στην Ισραηλινή ε, κυβέρνηση, αμυδρά μόνο. Ενδιαφέρεται για τις εντολές και παροτρύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ για τους οικισμούς και τα προϊόντα τους. Και μιλώ για, την, το Κοινοβούλιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ήδη το 2012 αλλά και το 2015 πιο πρόσφατα υποστήριξαν ότι ό,τι παράγεται στους οικισμούς δεν θα πρέπει να εισέλθει ε, χωρίς την ε, ε ξεκάθαρη σήμανση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προϊόντα από τους οικισμούς, επειδή ε, δεν αναγνωρίζονται από το Διεθνές Δίκαιο αυτοί οι οικισμοί, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ε, ο, θα θεωρείται ότι καλύπτονται ε, από την εμπορική συμφωνία ανάμεσα στο Ισραηλινό κράτος και την Παλαιστινιακή Αρχή. Σας ερωτώ λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακος των συνθήκων και δεν θα το αμφισβητήσετε. Και δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτά που κάνετε για τις διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί. Για ξέρω ότι είσαστε πραγματικά ε, αφοσιωμένοι σε αυτό. Ε, σας ερωτώ συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολήθηκε με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας για την σήμανση, την ετικετοθεσία αυτών των προϊόντων, κάνατε μελέτες, τι ξέρουμε, υπάρχουν στοιχεία. Εγώ ξέρω στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, ε, μπορεί ε, να αναγοράσει κάποιος κρασί από τους οικισμούς και αυτό αντιβαίνει ε, στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη ερώτηση και θα είναι πιο σύντομη. Ξέρετε ότι στην ε, Παλαιστίνη είτε μιλάμε για παιδότοπους, για σχολεία, για, για το δεξαμενές, διάφορα πράγματα καταστρέφονται από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει ε, αποζημίωση για αυτές τις καταστροφές, γιατί η Ένωση χρηματοδότησε αυτά τα προγράμματα. Και ε, γιατί δεν παρακρατούμε απλώς ποσά που στα πλαίσια των διμερών ανταλλαγών ε, διοχετεύουμε στο Ισραήλ. Γιατί δεν παρακρατούμε αυτά τα ποσά που αντιστοιχούν στην αποζημίωση αυτών των καταστροφών. Και κύριε Ντιμό, ε, μία σύντομη ερώτηση. Ο κύριος Λογάν Φαμπιούς, που ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών στη Γαλλία, είχε πει πως το θέμα της αναγνώρισης ε, του κράτους Παλαιστινής ε, θα συνδεθεί άμεσα με την ε, συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και την ενευτική διαδικασία του Ισραήλ. Δηλαδή, στο σενάριο που το Ισραήλ δεν θα δεχόταν να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αυτό ήταν το θέμα, ε, προτίθεται η Γαλλία να συνεχίσει ε, τη γραμμή ε, και να κρατήσει την υπόσχεση του Λογάν Φαβιούς που ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών τότε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντάκτουσον. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Η πρώτη απευθύνεται στον κύριο Βιμούν. Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Κέντρο για την ε, κοινή γνώμη μόνο ε, των τρίτων Παλαιστινίων υποστηρίζει την κυβέρνησή τους ε, που κυρώνει την γαλλική πρωτοβουλία το 35% λέει ότι η γαλλική πρωτοβουλία σέβεται τις απαιτήσεις των Παλαιστινίων. Σε σχέση με αυτό τα αρνητικά στοιχεία, αυτή η έλλειψη στήριξη που υπάρχει και από τι δύο πλευρέ, δηλαδή. Πώ μπορείτε να συνεχίσετε στην πρόθεση αυτή τη πρωτοβουλία. Δεύτερη ερώτηση για τον κύριο Τζεντιλίνη. Ο πρόεδρο Μαχμούτα Μπά έχει πολλά και σαρνηθεί να ξεκινήσει εκ νέου τις διμερείς διαπραγματευτικές διαδικασίες με το Ισραήλ, ακόμη και αν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό τον κάλεσε να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις χωρίς προαπαιτούμενα ο κύριος Νιτανιάχου επίσης εξέφρασε βούληση, τη βούλησή του να πάει στη Ραμάλα και να απευθυνθεί στο Παλαιστινιακό Κοινοβούλιο και επίσης κάλεσε τον κύριο Αμπάς να απευθυνθεί στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Με ποιο τρόπο, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν, ως ο μεγαλύτερος δωρητής κονδυλίων στην Παλαιστινιακή Αρχή, πιέζει την Παλαιστινική ηγεσία να επιστρέψει αμελητή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Φρόιντ. Ευχαριστώ πολύ. Χτες ε, το βράδυ είχαμε ένα πολύ καλό διπλό με την ομάδα νέων ηγετών από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ και αυτό που θα μπορούσαμε να αισθανθούμε σε καθαρίνο το ακόμη και αν βρίσκονται στην ίδια αίθουσα τους ε, χωρίζουν ε, ωκεανοί και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση είναι το πρώτο ζήτημα όπως ε, είπε ο καθηγητής. Θα ήθελα όμως να θέσω μία ερώτηση για δύο Αμερικανούς Προέδρους και οι δύο δεν είναι ο Τζίμι Κάρτερ ήταν στο παρελθόν ε, και έγραψε σήμερα στο New York Times και ζήτησε από τη σημερινή κυβέρνηση, την απερχόμενη κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Έτσι όπως έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες. Και αναρωτιέμαι αν ε, ο Λένε κάποιος άλλος θα ήθελε να το σχολιάσει αυτό και αν ε, κάτι τέτοιο είναι μια εφικτή οδός για τις επόμενες εβδομάδες μέχρι να αναλάβει τον Ντόναλτ Τραμπ. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον Ντόναλτ Τραμπ ε, και τις πολιτικές του για τη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτόν τελεία. Όμως, βασικά τι είπε ότι είναι καταπληκτικός ο λαός του Ισραήλ, τους συνάντησα όλους, είναι τέλεια η χώρα του Ισραήλ, όμως πέρα αυτού δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνάγουμε κάτι άλλο από τις δηλώσεις του. Όμως, στη συνέντευξη με τους New York Times είπε ότι ο Τζέρος Κούστνερ, ο γαμπρός του, θα είναι, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά θα είναι και εξαιρετικός άνθρωπος αν αναλάβει να εργαστεί για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και αναρωτιέμαι αν πρόκειται για μια ακόμη παράξενη ιδέα που εκφράζει που και που ο κύριος Τραμπ και αν έχει ουσιαστικά κάποια εγκυρότητα. Έχετε κάποιες ιδέες σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βανόρτεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι προλαλήσαντες αναφερθήκαν στην έλλειψη εστίασης ε, από την πλευρά των ΗΠΑ με την αλλαγή της Προεδρίας, όμως έχουμε και το ίδιο πρόβλημα αλλού. Και στη Γαλλία αυτή τη στιγμή έχουμε στο μέλλον προεδρικές εκλογές και μπορεί να υπάρχει αλλαγή της κυβέρνησης. Δεν ξέρω λοιπόν αν η Γαλλία θα συνεχίζει να επικεντρώνεται σε όλα αυτά περισσότερο από άλλους. Και πρέπει να αναρωτηθούμε, θέλουμε να συνεχίσουμε να εμπλεκόμαστε σε μάτες προσπάθειες ή θέλουμε να είμαστε ελπιδοφόροι. Και σε αντίθεση πώς εξέφρασαν κάποιοι συνάδελφοι, εγώ μπορώ να πω ότι δεν ξέρω κάποια χώρα που να θέλει ειρήνη περισσότερο από το Ισραήλ, ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια και ο Νετανιάχου έχει δεσμευτεί για τη λίστα των δύο κρατών. Α το έχουμε αυτό κατά νου. Οι Ισραηλοί έφυγαν από τη Γάζα και η Γάζα τώρα είναι στα χέρια μια τρομοκρατική οργάνωση. Έτσι λοιπόν ο λαό τη Γάζα δεν έχει καμία ελευθερία υπό τον έλεγχο τη Χαμά. Έχετε κατά νου ότι το Ισραήλ από την ίδρυσή του είναι ένα έθνο υπό Πριν από 69 χρόνια ξεκίνησε η επίθεση και είναι υποσυνεχή η επίθεση. Είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη χώρα, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Και τώρα, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης προσπαθεί απελπισμένα ε, ουσιαστικά να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην παγκοσμία σκηνή. Όμως εγώ θα πρότεινα, αντί αυτού, και θα αναφερθώ στο ΣΥΠΑ να χρησιμοποιήσει όποια μόχλευση έχει για να προσπαθήσει να αλλάξουν οι Παλαιστίνοι. Εμείς ε, είμαστε οι μεγαλύτεροι οικονομικοί υποστηρικτές των Παλαιστινίων. Και τι παίρνουμε σαν αντάλλαγμα γι' αυτό. Ποια πολιτική μόχλευση έχουμε επάνω τους. Καμία. Δεν βλέπουμε καμία πρόοδρο θα πρέπει να τους ξαναβάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αντί να κάνουμε μεγάλες χειρονομίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μικρότερα πράγματα. Παραδείγματο χάρη, βελτίωση σε ό,τι αφορά τη διαλευσή των συνόρων μεταξύ Δυτικής Όχθης και Γάζας. Και τι θα πρέπει να γίνει μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινιακών αρχών. Και θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλά πρακτικά έργα που θα μπορούσε να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να προκαλεί ουσιαστικά ψευδεστήσεις ε, σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με το θέμα της αναγνώρισης και ξέρουμε ότι η μόνη λύση που θα προκύψει είναι μέσω διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Και πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας να βοηθήσουμε και να μην κάνουμε αυτή την προοπτική ακόμη πιο μακρινή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Βάιντελ. Ευχαριστώ πολύ. Φοβάμαι ότι οι ομιλητές μετά από αυτή τη συζήτηση κατάλαβαν ε, ότι θα πρέπει να ακούσουν γιατί δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαρκματίσει κανένα ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθετες και βασικά μιλάμε δύο γλώσσες. Δεν πρόκειται περί της αναγνώρισης του Ισραήλ τις εγγυήσει και την πεποίθηση ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα ύπαρξης και να είναι ασφαλή, ασφαλές στα σύνορά του και την καταδίκη οποιοδήποτε θέλει να καταστρέψει αυτή τη χώρα. Χρειάζεται δηλαδή αυτή η καταδίκη και ήδη είναι κάτι ανεφεσβήτητο στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να δώσουμε μία όθηση σε αυτή τη διαδικασία η οποία είναι διαδικασία μόνο στα λόγια και είναι ειρήνη στα χαρτιά γιατί δεν υπάρχει καμία ειρήνη. Θα προσπαθήσω να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Είναι ενδιαφέρον που συζητάμε για τις Ισραηλο-Παλαιστινικές σχέσεις και το γεγονός ότι η λύση δύο κρατών γίνεται φάτα με κάθε μέρα που περνά δεν μιλάμε για τα μέσα που είναι ρεαλιστικά και διαθέσιμα και που η Ευρώπη θα μπορούσε ουσιαστικά να παίξει και ένα ρόλο, όπως είπε και ο καθηγητής πριν. Καταρχήν έχουμε την Γαλλική Πρωτοβουλία, έχουμε την Αραβική Ρηρευτική Πρωτοβουλία και υπάρχει και το Διεθνές Δίκαιο. Και τα μέσα που μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Αν σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο, αν εμένουμε στο διεθνές δίκαιο, γίνεται προφανές ότι το Ισραήλ δεν ε, είναι μόνο δημοκρατική χώρα της περιοχής, αλλά είναι και μια χώρα ότι παραβιάζονται οι δημοκρατικοί κανόνες και μάλιστα σοβαρά από την βασική μεταχείριση των άλλων των πληστινιών μέχρι τα 800 παιδιά που κρατούνται στη φυλακή μέχρι τους πάνω από 5.000 κρατούμενους υπό την απαράδεκτη συνθήκη της διοικητικής κράτησης βουλευτές είναι στη φυλακή κτλ. Ας μιλήσουμε λοιπόν ξεκάθαρα. Μπορείς να είσαι φίλος του Ισραήλ και να θέτεις αυτά τα ζητήματα διαφορετικά. Δεν θα κάνουμε καμία διαφορά. Σήμερα έλαβα μια ενημέρωση που θα σας κοινοποιήσω. Σε μία επιστολή στην κυρία Μογκερίνη, μία ομάδα μη κυβερνητικών οργανώσεων προσπαθεί να χρηστεί στην προσοχή μας ότι πέρσι το Μάιο ένα project ε, αφορά τον νόμο ξεκίνησε και υποστηρίχθηκε με ευρωπαϊκά χρήματα και αφορά την εναρμόνιση και ανταλλαγή τεχνικών ανάκρισης μεταξύ των διάφορων χωρών για να εντοπιστούν οι νέες προκλήσεις ε, της διεθνούς εγκληματικότητας. Συντονίζεται αυτό το project ε, από το Ισραηλινό Πανεπιστήμιο και συμμετέχει και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης Πορτογαλίας, η Χωροφυλακή της Ισπανίας κτλ. Και αυτό το έργο, αυτό το project, μιλά για τον εαυτό του. Γιατί οι ανακριτικές τεχνικές στο Ισραήλ, κάτι έχουμε ακούσει γι' αυτό και οι Παλαιστίνοι ξέρουν ακόμα περισσότερα. Πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε λοιπόν με τέτοιους όρους σε τέτοια project και ουσιαστικά να συνεχίζουμε τη δουλειά μας ως συνήθως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Λόπεθ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση ότι ε, η κατάσταση είναι παγωμένη, αυτή η σύραξη έχει πραγματικά εδραιωθεί και δεν απασχολεί και τόσο. Δεν γίνεται τίποτα από την διεθνή κοινότητα γι' αυτό. Οι βασικοί εμπλεκόμενοι δεν θέλουν να αναλάβουν το κόστος που θα είχε μια διαπραγματεύση για να επιτευχθεί λύση. Ας θυμηθούμε ότι από το 2006 δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική αλλαγή. Από το 2006 είχαμε την πρωτοβουλία του ε, Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Κέρι, αλλά δεν, ε, δεν ε, είχε κανένα αποτέλεσμα. Ερωτήσεις λοιπόν. πώς θα τους πείσουμε να κατέβουν στις διαπραγματεύσεις εφόσον έχουν τόσες διαφορετικές προϋποθέσεις. Άλλοι θέλουν ε, πολυμερή διάσκεψη ενώ το Ισραήλ θέλει διμερείς ή με τις ΗΠΑ. Οι Παλαιστίνοι αναφέρουν μια σειρά από προϋποθέσεις, σύνορα, κατοχή. Οι Ισραηλοί λένε όχι, να μην υπάρχουν απριόρι για τη διαπραγμάτευση. Πώς, τι θα κάνουμε. Γιατί έχουμε πέσει σε τείχο τα τελευταία χρόνια. Όλοι λέμε ότι πώς θα ενισχύσουμε την επιρροή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα ασκήσει επιρροή. Παρά τις διαφορετικές απόψεις, όλοι οι, όλοι οι βουλευτές είπαν ότι θα θέλαμε η Ένωση να έχει περισσότερη επιρροή. Πώς θα το κάνει, πώς. Έχουμε μια σειρά μέσα, την αγορά, για το Ισραήλ, την αγορά μας για το Ισραήλ και όλες ε, τις χρηματοδοτήσεις που δίνουμε στην ε, Παλαιστινική Αρχή. Αλλά πώς θα έχουμε περισσότερη επιρροή. Τρίτον, ε, η ερώτησή μου για τα δύο κράτη είναι νομίζετε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή που δεν θα είναι πια για πρακτικούς λόγους αδύνατο να υπάρχουν δύο κράτη. Εάν ο κατακαιρματισμό ε, των ε, παλαιστινιακών εδαφών, η πολιτική καμένης γης, οι δημογραφικές αλλαγέ, οι επικισμοί, αν όλα αυτά θα μας οδηγήσουν κάποια στιγμή που δεν θα είναι πια ε, πρακτικά δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Παρά το ότι όλοι και εγώ συμμερίζομαι τη λύση των δύο κρατών. Και τέλος, Υπάρχουν κάποια στοιχεία που λένε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια ε, συμφιλίωση μεταξύ των διαφόρων παλαιστινιακών δυνάμεων. Εάν γίνει κάτι τέτοιο θα βοηθήσει τη διαδικασία ειρήνευση. Πρόεδρος. Ο Κρίστιαν Πρέντα. Ευχαριστώ. Μα τα έχουμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα ήθελα να πω τα θέματα αυτά και είναι σαν να ξανακούν τα ίδια η ομάδα μας πρότεινε να συζητήσουμε πρώτα απ' όλα στην ΑΦΕ το θέμα αυτό. Εγώ πάντα εκφράζω ιδιαίτερη απογοήτευση βλέποντας ότι από τη μία ορισμένοι συνάδελφοι εκφράζονται κατά των απευθείας διαπραγματεύσεων. Εάν θέλουμε κάτι να επιτύχουμε, πρέπει να ζητήσουμε να γίνουν απευθεία διαπραγματεύσει μεταξύ των δύο πλευρών χωρί προποθέσει. Γιατί αλλιώ θα έχουμε όλο αυτό τον κατάλογο από διακηρύξει όπου ο ένα καταδικάζει τον άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα όχι, μάλλον όλοι καταδικάζουμε έναν από τις, μία από τις δυνάμεις, είπε ο κύριος Πρέντα. Και τώρα να απαντήσουν οι ομιλητές μας. Λοιπόν, βάζω το χρονόμετρο. 5 έως 7 λεπτά ο καθένας. Με την αντίστροφη σειρά. Ο δόκτωρ Μπεν Μέιρ πρώτος. Μετά ο κύριος Βήμο και μετά ο κύριος Τζεντιλίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ρωτηθήκαμε, μπορούμε να προβλέψουμε την πολιτική Τραμπ. Όχι, να μην κάνουμε προβλέψεις θα έλεγα όσον αφορά την σύραξη. Μπορώ να σας πω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να στηρίζει το κράτος του Ισραήλ με βάση όσα γνωρίζω. Πιστεύει σε λύση δύο κρατών, αλλά ακόμη δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα, καμία στρατηγική από πλευράς ε, της νέας κυβέρνησής του για να εκινήσει αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό λέω ότι επειδή είναι απαραίτητες οι Ηνωμένε Πολιτείε για την επίλυση, γι' αυτό προτείνω να λάβουμε υπόψη ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν πρόκειται τώρα να εμπλακεί για αυτό το θέμα. Γι' αυτό πρέπει να τους δώσουμε, να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα να προλιάνουμε το έδαφο. Όχι να αντικαταστήσουμε τι ΗΠΑ, αλλά σε 1,5-2 χρόνο λοιπόν οι δύο πλευρέ να είναι πολύ πιο διατεθειμένε να αρχίσουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο, τι παραχωρήσει πρέπει να κάνουν, ούτω ώστε ενδεχομένω να καταλήξουν να τι κάνουν. Τώρα μια διάκριση που πρέπει να κάνουμε. Το Ισραήλ ω χώρα και η κυβέρνηση. Πρέπει να τα, να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Συμφωνώ με τον κύριο Βημού ε, όλες οι δημοσκοπήσεις ε, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των πληθυσμών στηρίζουν τη λύση των δύο κρατών. Οι κυβερνήσει είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι, κάποιο με ρώτησε, ναι, βεβαίως μπορώ να πω, έχω το θάρρος να πω, ότι η σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση και η σημερινή Παλαιστινική Αρχή μπορούν να κάνουν τι αναγκαίε για επίλυση. Εάν ο κύριος Νετανιάχου κάνει οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια, η κυβέρνησή του θα διαλυθεί την ίδια μέρα. Διότι είναι κυβέρνηση συνασπισμού και ορισμένοι συμμετέχοντες καλούν για προσάρτηση της Γάζας, ε, το, συγγνώμη, της Δυτικής Όχθης. Και τώρα, η Χαμάς θα πρέπει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ε, ειρηνευτική διαδικασία μόνο με την Παλαιστινική Αρχή. Πρέπει να συμμετάσχει και η Χαμά. Παρά τι δημόσιε διακηρύξει που θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ, η Χαμά επίση γνωρίζει και το ξέρω από πρώτο χέρι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να καταστραφεί και ότι πρέπει να βρεθεί τρόπο για να συνεπάρξουν με το Ισραήλ. Και γι' αυτό, αυτό που σα λέω σήμερα είναι ότι η αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία του δίνει μια ε, οδό διεξόδου. Οι χώρες που μπορούν να επηρεάσουν τη Χαμάς, Τουρκία, Κατάρ, μπορούν να αρχίσουν ένα διάλογο με τη Χαμάς για να την κάνουν να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Η Χαμάς είναι διατεθειμένη, αλλά πρέπει να της δοθεί μια διέξοδο. Η Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία μπορεί να της την παράσχει. Η συζήτηση για το θέμα αυτό μπορεί να γίνει ε, μέχρι για εβδομάδες, αλλά η αρχή αυτή ισχύει. Όσοι είναι σε επαφή με το Κατάρ, την Τουρκία και τη Χαμάς λαμβάνουν τα ίδια μηνύματα. Είναι απολύτως εφικτό κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε την καταμέτρηση όλων των λαθών και αποτυχιών και των δύο πλευρών στο παρελθόν. Κανένας δεν προτείνει ότι το Ισραήλ είναι άμομο. Ούτε οι Παλαιστίνοι ότι ήσαν άμομοι και οι δύο έκαναν τραγικά σφάλματα τα τελευταία 50 χρόνια και συνεχίζουν να διαπράττουν τραγικά σφάλματα. Και προσπαθούμε, μπορούμε να πούμε, μπορούμε να αρχίσουμε να προσπαθούμε να πούμε ποιο φταίει περισσότερο. Όμω ε, κάτι είναι σαφέ. Η κατοχή δεν είναι βιώσιμη. Πρέπει κάποτε να λήξει. Και για το πώ θα λήξει είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία που ανέφερα προηγουμένω. Και εδώ έχουμε τη δυσχέρεια που πρέπει να την εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Ποιοι θα συμμετάσχουν στη Γαλλική Πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε διεθνής διάσκεψη, εάν δεν συμμετέχουν σε αυτή και το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, δεν λέω ότι θα είναι εντελώ ε, χάσιμο χρόνου, αλλά δεν θα έχει αποτελεσματικότητα. Πρέπει να συμμετέχουν και οι δύο αυτέ πλευρέ, εφόσον Ε, ξέρετε, ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να συμμετάσχει αν ε, θεωρήσει ότι θα πιεστεί υπερβολικά. Πρέπει να τους πούμε ότι αυτή η διάσκεψη πρέπει να καταλάβουν ότι θα είναι η εκκίνηση μιας νέας διαδικασίας. Διαδικασία συμφιλίωση. Δεν θα κάνουν ουσιώδε παραχωρήσει κατά τη διάρκεια τη διάσκεψη, αλλά μπορούν να έρθουν για να καταλάβουν ότι χρειαζόμαστε μια διαδικασία συμφιλίωση, ούτω ώστε οι δύο λαοί να έρθουν πιο κοντά ένα στον άλλον, να μετριαστεί η δυσπιστία, ε, η αίσθηση ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, ε, να σταματήσουν οι ψευδεστήσεις ότι μπορώ να επιτύχω το maximum των ε, βλέψεών μου. Ε, αλλιώς δεν θα έχει επιτυχία. Τώρα ο Ομπάμα, συγγνώμη, το ότι ο κύριος Κάρτερ ζήτησε από τον πρόεδρο Ομπάμα να αναγνωρίσει το Παλαιστινικό κράτος πριν αποχωρήσει, δεν νομίζω ότι είναι και καλή συμβουλή. Δεν θα αλλάξει τίποτα επί τόπου. στην ουσία θα ενισχύσει τους πιο ακραίους ε, στο Ισραήλ. Και δεν θα υπάρχει μηχανισμός ε, επιβολής αυτής της απόφασης. Και μετά θα μπει ο πρόεδρος Τραμπ στο Λευκό Οίκο και θα πει όχι, δεν ισχύει αυτό. Το να πει απλώς να κάνει μια διακήρυξη ο πρόεδρος Ομπάμα και να θεωρήσει ότι αυτό θα έχει μακροπρόθεσμη ε, επίδραση δεν νομίζω ότι ισχύει και είναι λάθος λοιπόν η πρόταση Κάρτερ. Δεν νομίζω ότι οι προσπάθειες ε, της Ένωση των Γάλλων ή κάποιου άλλου είναι άσκοπες. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε την κατάσταση όπως είναι τώρα. Πρέπει να υπάρξει κάποια δράση, κάποιες δραστηριότητες για να ε, σταματήσουμε τη δημιουργία νέων καταστάσεων επιτόπου που καθιστούν την κατάσταση, καθιστούν την κατάσταση όλο και περισσότερο μη αναστρέψιμη και οριστική και που καθιστούν την προοπτική ειρήνη ε, αδύνατη, σχεδόν αδύνατη. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία συμφιλίωσης για να επιβραδύνουμε, αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δημιουργία όλο και νέων καταστάσεων επιτόπου που θα καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε λύση, ιδιαίτερα την λύση των δύο κρατών. Να σταματήσω εδώ. Καλά, σταματάω λοιπόν. Θα σταματήσω γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε καθηγητά Μπριμέιρ. Κύριε Βήμου, δεν θα υπερβώ το χρόνο μου. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις για πρώτα απ' όλα για τη διάσκεψη. Και αν θες μετά στην Ισραηλινή κυβέρνηση ή όχι, ρωτήσατε εσείς κύριε Παρνιό αν δεν κάνω λάθος. Εξ αρχής ε, μας είπαν ότι διαφωνούν με την πρωτοβουλία μας και τώρα που μιλάνε για τη τελική διάσκεψη ε, δηλώνουν ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να συμμετάσχουν. Το σημειώνουμε φυσικά και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε αφενός να προχωρήσουμε με τη διάσκεψη για όπως σωστά είπε ο αφετέρου να έχουμε μια διάσκεψη όπου δεν θα αποκλειστεί κανείς γιατί αν απουσιάζει κάποια πλευρά θα δημιουργηθεί η αίσθηση ανισορροπίας. Προσπαθούμε να βρούμε ε, τον ορθότερο τρόπο για να προχωρήσουμε. Όπως είπε ο καθηγητής ε, Μπεν Μέιερ, αυτή η διάσκεψη δεν έχει ως στόχο να ασκήσει πίεση προς κάποια πλευρά και να γίνει μια αμφιλεγόμενη διάσκεψη. Να θυμίσω κάποια στοιχεία και κάποιες αρχές επί των οποίων ε, οικοδομήσαμε τη διάσκεψη δεν θέλουν να συμμετάσχουν, ναι. το να μας λένε ότι δεν ναι, συντρέχει ανάγκη να επαναλάβουμε αυτές τις αρχές, ενώ όμως ακολουθεί η λανθασμένη κατάρρυθμιση, η διαδικασία μας φαίνεται ότι είναι άτοπο. Και έχουμε την εντύπωση ότι ε, εκλείπει από την όλη εικόνα η, ε, ολένα και περισσότερο η λύση των δύο κρατών και αυτό μας ανησυχεί. Η υποστήριξη από την Παλαιστινιακή πλευρά. Μπορώ να σας πω πως ε, εάν υπάρχει ένας εταίρος στη διεθνή κοινότητα που υποστήριξε εξ αρχής τη Γαλλική Πρωτοβουλία είναι η Παλαιστίνη. Εξ αρχής ε, μας είπαν ότι είναι ο μόνος τρόπος, σας υποστηρίζουμε σε τέτοιο βαθμό που θα έλεγα ότι ίσως έχουν και υπερβολικές προσδοκίες από τη διάσκεψη. Και τα μηνύματα που παίρνουμε από την Παλαιστινιακή Αρχή και από τους ηγέτες των κοινοτήτων είναι ξεκάθαρα. Δεν υφίσταται καμία αμφισημία. Και θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε για το χρονισμό ο καθηγητής Μαέρ ότι ενδεχομένως καλύτερα να περιμένουμε και να αναβάλουμε προς το παρόν τη διάσκεψη. Δεν κρίνω ότι υπάρχει σωστή λύση. Αν δηλαδή περιμένουμε την ορκομοσία του Τραμπ ή όχι. Υπάρχουν υπέρ και κατά σε όλες τις περιπτώσεις. Να περιμένουμε λοιπόν και η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει αυτή τη γραμμή, διότι είναι σημαντικό να το θυμίσουμε. Εάν αναβάλουμε τη διάσκεψη και όπως είπε ο καθηγητής Μπεν Μάιρ, η νέα κυβέρνηση ζήτησε χρόνο ε, για να ε, σκεφτεί την όλη διαδικασία, δεν θα είναι ένας μήνας. Θα παραταθεί πολύ η διαδικασία. Ο καθηγητής Μάιρ είπε να προλιάνουμε το έδαφος ε, τα επόμενα δύο χρόνια για να έχουμε την ε, συμφιλίωση στο πέρας της διαδικασίας. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει αμελητή να ξεκινήσουμε. Τρίτο σημείο για αναγνώριση. Εάν ε, αποτύχει η πρωτοβουλία τότε θα εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Και αφήνοντας την επι... όλη επιχειρηματολογία, μπορώ να σας πω ότι ανάμεσα από αυτή την σύνδεση των δύο στοιχείων ναι, προέκυψε ότι πολλοί εταίροι μας ίσως είχαν ενδιασμούς. Δηλαδή να ε, συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την πρωτοβουλία που ενδεχομένως ε, ε, στο τέλος να ανοίξει το δρόμο της αναγνώρισης. Και γι' αυτό αποφασίζαμε να το αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν. Και το θέμα της αναγνώρισης ή μη αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, έχουμε πει, είναι θέμα εθνικό, θέμα κυριαρχίας για τη γαλλική κυβέρνηση. Και άρα θα πρέπει να προσέξουμε τη σύνδεσή του με μια διάσκεψη όπου επιθυμούμε τη μέγιστη, την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Και αν τελευταίο σημείο και πρόεδρε θα σταματήσω μετά. Άκουσα από διάφορε πλευρέ ότι θα, θα πρέπει να διεθνοποιήσουμε τη διαδικασία και θα πρέπει να μιλάμε για άμεσε διαπραγματεύσει. Ε, θα ήθελα να ε, διαλύσω αυτή την αμφιβολία που υπάρχει και την ε, παρανόηση. Φυσικά είμαστε ε, υπέρ των άμεσων επαφών. Να καθίσουν στο δύο τραπέζι όλοι. Αυτή είναι τον όνων κάνει προπόθεση για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι ασύμβατες οι δύο γραμμές. Το αντίθετο είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Είναι σημαντικό να το πούμε σε σχέση με την διεθνοποίηση ε, της διαδικασίας, επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο καθηγητής Εμπενμερή για την συνύπαρξη. Είναι ένα δεδομένο και πρέπει να το δεχτούμε. Το ίδιο ισχύει και για τη διεθνή διάσταση του ζητήματος. Η αρρωγή, παραδείγματο χάρη. Ποιο βοηθάει του Παλαιστινίου, ποιο βοηθάει του Ισραηλινού με ερευνητικά προγράμματα, με εμπορικά προγράμματα, η σύσσωμη διεθνή κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, η Ρωσία κτλ. Είναι προ συμφέρον όλων, άμεσο συμφέρον όλων να εγκαθιδρυθεί η ειρήνη γιατί ε, το θέμα είναι και η δική μας σταθερότητα, η δική μας ασφάλεια. Το να προσπαθήσουμε να, να ε, διαχωρίσουμε αυτά που συμβαίνουν στη διεθνή κοινότητα και αυτά που συμβαίνουν επί τόπου, είναι ε, αντίθετο προς την πραγματικότητα που παρατηρούμε επί τόπου, κατά τη γνώμη μου. Εδώ και θα σταματήσω. Ευχαριστούμε κύριε Ντίμο. Ο κύριο Τζεντιλίνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Θα προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω. Καταρχήν, για το ρόλο των ε, Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη ΣΥΠΑ. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις ε, που έθεσαν αυτή την αντίφαση. Αναφερθήκατε και εσείς, Πρόεδρε, για να είμαι σαφής. Τι ήθελα να πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι είναι πιο ισχυρή αν βρέσει από κοινού με το διεθνή της εταίρο. Νομίζω αυτό είναι το θέμα. Επίσης είναι πιο ισχυρή σε ό,τι φορά τη μόχλευση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που τέθηκε. Νομίζω ότι ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Μπορεί να φαίνεται προφανές, αλλά δεν είναι. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το έχουμε κατά νου. Γι' αυτό έχουμε επενδύσει πολύ σε αυτό το έργο με το κουαρτέτο και τους εταίρους μας εκεί. Και γι' αυτό πάντοτε εργαζόμαστε σκληρά βάση και τον ε, τι λένε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι θέσεις μας κτλ. Για την Αμερικανική κυβέρνηση, όπως ε, υπόθηκε, ήμουν και στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, συμφωνώ με όσα υπόθηκαν, αλλά ένα πράγμα που είναι βέβαιο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενδιαφέρον να εμπλακεί στη διαδικασία. Γιατί από κοινού είμαστε ισχυρότεροι και μπορούμε να δώσουμε όθηση στα θέματα αυτά. Εδώ βλέπω ότι γίνεται επιτόπου. Πολύ καλά να έχουμε δύο πλευρές να προσπαθούν ε, να βρουν ε, το χώρο τους μεταξύ των διάφορων εταίρων, αλλά ενωμένοι είμαστε δυνατότεροι και ίσως μπορούμε και να τα καταφέρουμε. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα για άλλο σύνολο ερωτήσεων το θέμα της προθυμίας των δύο πλευρών να διαπραγματευτούν. Δηλαδή μια πλευρά προσφέρει δυνατότητα συνάντησης, η άλλη όχι και ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό. Θέλω να είμαι σαφής και να τονίσω κάποια θέματα που ήδη αναφέρθηκαν. Κανείς θεωρώ ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις δύο πλευρές, τα δύο μέρη. Σε αυτό το παιχνίδι Κανείς δεν μπορεί λοιπόν να αντικαταστήσει τα δύο μέρη, ούτε τις άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές, αποτελεί και μια σαφή βάση για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στον τομέα αυτό. Βέβαια, ένας συνοδευτικός μηχανισμός είναι πάντοτε σημαντικός και νομίζω ότι η φιλοδοξία θα ήταν να έχουμε αυτό τον βοηθητικό μηχανισμό, καταρχήν με τους περιφερειακούς εταίρους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και τους άλλους παίκτες. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ενωμένο διεθνές μέτωπο. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι δεν είναι θέμα μόχλευσης, αλλά θέμα πολιτικής βούλησης. Και αυτό είπα. Πρόκειται για πολιτική βούληση σε σχέση με το τι θέλουμε να κάνουμε, με το πώς προχωρούμε. Όπω υπόθηκε, δεν νομίζω ότι πρέπει να επαναφεύρουμε τον τροχό. Κάποια από αυτά τα βήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να ξαναδημιουργηθούν οι συνθήκε ε, για ουσιαστικέ συνομιλίε, ε, όταν είναι κατάλληλο το πλήρωμα του χρόνου, υπάρχουν και συμφωνώ όμω, υπόθηκαν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα μικρά πρακτικά βήματα, συγκεκριμένα βήματα, γιατί και αυτό είναι προφανέ να το λέει κανεί, αλλά σε ένα τέτοιο ζήτημα νομίζω ότι είναι φυσικό να πηγαίνουμε από τα πιο εύκολα στα πιο δύσκολα ζητήματα. Όλοι συμφωνούμε από αυτού, αλλά νομίζω ότι εδώ το θέμα κλειδί είναι η πολιτική βούληση. Επίσης συμφωνώ με όσους έθεσαν το θέμα της Γάζας. Είναι σημαντικό ζήτημα. Δεν συζητάμε ποτέ αρκετά για τη σημασία της Γάζας, όμως και πάλι στην έκθεση του κορτέτου και στις συστάσεις υπάρχει αρκετός χώρος που αφιερώνεται για το θέμα αυτό, την, ε, το πρόβλημα του αποκλεισμού, της ε, στρατιωτικής ε, διαδικασίας που ακολουθείται εκεί, την ανάγκη να υποστηριχθεί ο πληθυσμός και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ενεργή μέσω των δικών της διάβλων και φυσικά υπάρχει και έσχατη ανάγκη επανασυμφιλίωσης γιατί σύμφωνα με τις αρχές του κουαρτέτου και τις αρχές της πιλότης ε, ε, παραμένει το θέμα της συμφιλίωσης ένα πολύ σημαντικό. Επίσης ε, τέθηκε και το θέμα των επικισμών και το θέμα των καταστροφών. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο ε, που αφορά την ε, τάση αυτή στη δυτική όχθη. Ηνωμένοι είμαστε ισχυρότεροι και δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τη σημασία του να έχουμε μια κοινή αξιολόγηση επί των ε, τάσεων και μια κοινή συνταγή για το πώς θα προχωρήσουμε προς τα μπρος. Θα είναι εύκολο? Όχι. Δεν είναι εύκολο και το βλέπουμε καθημερινά, Όμω το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να, ε, να το κάνει αυτό, γιατί η αντιπροσωπεία μας στο κύριο Δημήμα έχει ένα διορθωτικό διάλογο, τρωμένο διάλογο, συγγνώμη, με το Τελαβίβ, με το Ισραήλ, στο θέμα αυτό. Και είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την πίεση. Για ένα άλλο σημαντικό θέμα που αναφέρθηκε για την ε, ένδειξη είναι σαφή η απάντηση. Και για να μην μακρηγορώ, είναι πολύ σημαντικό πάντοτε να διακρίνουμε τι είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και τι, είναι, τι εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, κυρίω ό,τι αφορά την εφαρμογή κάποιων πραγμάτων. Κοιτάξτε, τώρα για αυτό το project που αναφέρεται για την κατάρτιση, ε, σε νομικά ζητήματα δεν είμαι αρμόδιος και δεν μπορώ να απαντήσω. Όμως ευχαριστώ να επανέλθω διμερώς αυτή διαβουλευτώ με τον συναδελφό μου. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στο πάνελ και όλους ε, όσους ε, θέσατε ερωτήσεις και κάνατε σχόλια. Μπορούμε λοιπόν εδώ να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σας ευχαριστώ. colleagues, um, uh, Συνάδελφοι, τώρα θα συζητήσουμε την έκθεση για την Βοσνία Ζεγοβίνη. Και δίνω το λόγο Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Πρέντα. Που είναι και ο Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Λοιπόν, έχουμε την έκθεση για την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μετά την έκθεση που πριν από τρεις εβδομάδες υπέβαλε η Κομισιόν. Το κείμενο υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Είμαι πεπισμένος ότι θα με συγχωρήσουν γι' αυτό οι συνάδελφοι. Επειδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έκθεση αυτή πιο γρήγορα από ό,τι πέρυσι για να ψηφίσουμε τον προσεχή Φεβρουάριο στην Ολομέλεια. Το 2017 είναι σημαντική χρονιά για τη χώρα, γιατί οι αρχές του Σαράγεβο ελπίζουν η χώρα να αποκτήσει πριν το τέλος του 2017 καθεστώς υποψηφίου χώρας. Επιπλέον, αντίθετα από φέτος και το 2018 το 2017 δεν ε, υπάρχουν εκλογές. Πρέπει να αποφεληθούμε. Γιατί ξέρουμε ότι πολύ συχνά για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη οι εκλογικές διαδικασίες ε, σημαίνουν ότι όλα σταματάνε και όλοι εργάζονται μόνο για τις εκλογές. Η έκθεση λοιπόν ε, της Ευρωπαϊκής Επιτρόπης είναι η δεύτερη θετική έκθεση για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι είναι συνέχεια της έκθεσης ε, του 16. Είχαμε το πρώτο πρωτόκολλο που είναι η προσαρμογή μετά από την ε, ένταξη της ε, Κροατίας που περιμένουμε να υπογραφεί το Δεκέμβριο. Αυτή είναι η δεύτερη καλή είδηση. Κατόπιν έχουμε συμφωνία για την ε, ολοκλήρωση του μηχανισμού συντονισμού που καταφέραμε να ε, ολοκληρωθεί στις 23 Αυγούστου μετά από χρόνια ακινησίες. Λήφθησαν πολλές πρωτοβουλίες για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ή συγγνώμη οι μεταρρυθμίσεις και τελικά υπάρχει, υπήρξε στις 20 Σεπτεμβρίου συνένεση στο Συμβούλιο για να συζητηθεί η ε, αίτηση ένταξης της Κροατίας και το Συμβούλιο ε, επεφόρτησε την Κομισιόν να κάνει μια έκθεση και θα έχουμε λοιπόν την ε, έχουμε το ρετματολόγιο της Κομισιόν και αρχές Νοεμβρίου λέει ο μιλητής, ο κύριος Χάν θα πάει στο Σαράγεβο για μια ε, επίσημη διαδικασία. Για τη Βοσνία Ζεγοβίνη είναι μέγιστη σημασία σε αυτή η εξέλιξη. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τις αρχές της χώρας να συνεργαστούν με συντονισμένο τρόπο γιατί οι ερωτήσεις στο ρηματολόγιο πρέπει να είναι μία σε κάθε οι απαντήσει μάλλον, μία σε κάθε ερώτηση. Και ελπίζω να μην λάβουμε τι απαντήσει γιατί δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ του. Γιατί σε κάθε ερώτηση λοιπόν του ερωτηματολογίου χρειάζεται μία απάντηση. Πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουν μεταξύ του. Και υπογραμμίζω ότι θα του τεθούν και συμπληρωματικέ ερωτήσει. Η διαδικασία θα συνοδευτεί από αποστολέ επιτόπου. Όλοι θα έχουν δυνατότητα να εκφραστούν λοιπόν. Αλλά οι απαντήσει στα ερωτήματα πρέπει να είναι ενιαίες. Δεν μπορούμε να λάβουμε απαντήσεις ανά εθνότητα, ανά πολιτικό κόμμα, ανά δεν ξέρω εγώ τι φιλοδοξία του κάθε ηγέτη. Πρέπει οπωσδήποτε βεβαίως να χαιρετήσουμε την πρόοδο που σημειώθηκε για την εφαρμογή του θεματολογίου για τις μεταρρυθμίσεις. Έχουν δεσμευτεί να κάνουν κοινωνικονομικές περίπλοκες μεταρρυθμίσεις οι αρχές της χώρας και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πορεία. Ελπίζουμε πάντα ότι ότι θα έχουμε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Γιατί απλώς ε, η εντύπωση που θα τους δοθεί είναι ότι υπάρχουν μεταρρυθμίσεις αλλά δεν έχουν επιπτώσεις για την καθημερινή ζωή των πολιτών, για την κοινωνία. Δύο λοιπόν πρέπει να υπογραμμιστούν, δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα οι προσπάθειες για τις μεταρρυθμίσεις πρέπει να περάσουν πάνω από τις εθνικές και πολιτικές διαφορές. Γιατί είδαμε την περίοδο Φεβρουαρίου-Αυγούστου πολλές διαφορές και διχόνοιες. Και επίσης οι διακηρύξεις περί ευρωπαϊκής πορείας πρέπει να μεταφραστούν σε πρόοδο για το κράτος δικαίου, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Και επίσης ε, πρέπει να υπάρξει εκβάθρον μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκηση. Εάν δεν υπάρχει κράτο δικαίου που να λειτουργεί, εάν δεν αντιμετωπιστεί η διαφθορά που έχει κατασταθεί και εντό των πολιτικών κομμάτων, δεν έχουν έννοια όλα αυτά. Τα ίδια τα πολιτικά κόμματα πρέπει να καθαρίσουν το σπίτι τους, τη χώρα τους, για να απομακρυνθούν από την πολιτική διεφθαρμένη. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός συντονισμού, καλό αυτό, αλλά ανεπαρκές. Πρέπει και να λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα. Ο ρόλος της διεύθυνσης για την ευρωπαϊκή ένταξη πρέπει να ενισχυθεί. Έχει μερικά πολύ καλά στελέχη, αλλά πρέπει να τα βοηθήσουμε. Κάτι άλλο σημαντικό που το έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου και είμαι εδώ δίπλα στο φίλο μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Συντονισμού. Ακόμη δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί λόγω διαφόρων ε, πολιτικών βλέψεων υπερβολικών. Και επανειλημμένα το έχουμε τονίσει, το ξαναλέω, έναντι των ηγετών της χώρας, ότι πρέπει να κατανοήσουν ότι είναι ένα εργαλείο που θα του βοηθήσει. Δεν είναι ένα φόρουμ που θα λαμβάνει αποφάσεις, αλλά πρέπει να μπορούμε να έχουμε ανταλλαγές απόψεων με τους ε, βουλευτές της χώρας. Εμείς οι ευρωβουλευτές το κάνουμε σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι η μόνη χώρα όπου δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα έχω δυνατότητα να το πω και στον πρόεδρο Μλάντεν Ιβανιτς που θα είναι εδώ αύριο γιατί η σερβική κοινότητα έχει ιδιαίτερη ευθύνη για το θέμα αυτό. Θα του το πω πολύ ανοιχτά. Καλά τα πήγανε οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολύ καλή διεξαγωγή, συγχαρητήρια στις αρχές. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν δύο επεισόδια. Ιδιαίτερα λυπηρά. Πρώτα απ' όλα στο Στολάτς όπου ένας ε, υποψήφιος άσκησε βία κατά του εκλογικού αντιπροσώπου που μπλόκαρε τη διαδικασία. Δεν μπορούσαν να ψηφίσουν εκεί οι άνθρωποι. Ανεβλήθησαν οι εκλογές και αυτό είναι απαράδεκτο. Και επίσης οι κάτοικοι του Μοστάρ δεν είχαν δυνατότητα να ψηφίσουν. Είμαστε εκεί τόπου ως αντιπροσωπεία ΑΦΕΤ. Είδαμε εκεί όλους τους ηθήνοντες, όλοι είπανε ναι, ναι, θα γίνει, θα γίνει και δεν έγινε τίποτα. Όπως εδώ και χρόνια. Δεν υπήρξαν εκλογές στο Μόσταρ. Και πόσο συμβολική είναι αυτή η χώρα, η πόλη για τη χώρα. Η καταπολέμηση της διαφθοράς, ήδη τα είπα, να προσθέσω ότι μια Πρόσφατη έρευνα της Transparency International δείχνει ότι 82% των πολιτών της χώρας θεωρούν ότι οι αρχές δεν αντιμετωπίζουν καλά ή όχι επαρκώς καλά την ε, διαφθορά. Άρα εφόσον ε, κάποιοι πολιτικοί γιατί είναι υπεύθυνοι θα πρέπει κάτι να κάνουν. Τώρα για τη δημόσια δίκηση. Υπάρχει υπερπολιτικοποίηση, αναποτελεσματικότητα, της διοίκησης. Λυπηρό αυτό, αλλά θέλουμε να τους ε, καλέσουμε να υπερβούν αυτές τις καθυστερήσεις. Σεβασμός του κράτους δικαίου. Είναι λυπηρό ότι πολλές αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου δεν εφαρμόζονται. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ακριβώς είπε ότι 93, 92 συγγνώμη, αποφάσεις έχουν μείνει νεκρογράμμα και μία ιδιαίτερα είναι πολύ ανησυχητική η απόφαση για την περίφημη πλέον υπόθεση του δημοψηφίσματος της 25 Σεπτεμβρίου που εργάνωσε ο Μίλο Αντόντιτς στην Σερβική Δημοκρατία αρνούμενος ανοιχτά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αρνώντας την παρά τις προσπάθειές μας παρά και τις προσπάθειες των φίλων στη Βοσνία Ζεγοβίνη, δεν ε, μπορέσαμε να πείσουμε τον κύριο Ντόντιτς ότι δεν είναι τρόπος αυτός. Γιατί προτιμάει να ακούει αυτά που του λέει ο κύριος Πούτιν. Δύο μέρες μετά το δημοψήφισμα πήγε και επισκέφθηκε τον Πούτιν για να πει από που ε, πρέπει να παίρνει εντολές. Δεν ενδιαφέρεται η Ρεπούμπλικα Σέρψκα, η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας Αζεγοβίνης για αυτά που τις λένε οι Βρυξέλλες, αλλά για αυτά που τις λέει η Μόσχα. Έτσι αγνώρισαν την απόφαση του ε, συνταγματικού δικαστηρίου. Αυτό το μήνυμα μας ήταν ο Ντόντιτς. Καταπολέμηση τώρα του οργανωμένου εγκλήματος. Χρειάζεται συντονισμός μεταξύ των αρμοδιών αρχών σε διάφορα επίπεδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμη περιμένουμε μια συνεπή στρατηγική για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Λοιπόν, προχωρώ. Ένα θέμα που ε, συνεχίζει να μας ανησυχεί και αναφέρεται σε κάθε της έκθεση είναι ότι η χώρα εξακολουθεί να μην σέβεται την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιατί δεν εφαρμόζει τις ε, επαφώσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις περιπτώσεις Ζένης, Ζήνης, Ζόντιτς και Πιλάφ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ξεχάσουν οι αρχές της χώρας αυτές τις αποφάσεις γιατί μπορούν να τις ξεχνάνε αυτοί, αλλά εμείς τους τις θυμίζουμε και περιμένουμε να τις εφαρμόσουν. Η κατάσταση των δημοσιογράφων και των μέσων πολύ ανησυχητική τους. Συναντήσαμε πρόσφατα διάφορες ενώσεις. Πολύ συχνά ε, ε, ασκούνται πιέσεις επί των δημοσιογράφων, αλλά δεν γίνονται έρευνες. Ακόμη και πράξεις βίας, βιοπραγίες. Αλλά δεν γίνονται έρευνες. Για τα οικονομικά θέματα, στις παραγράφους 21 και 22 της έκθεσής μου αναφέρομαι ιδιαίτερα ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η ανεργία και ιδιαίτερα η ανεργία των νέων. Αναμένουμε η κυβέρνηση κάτι να κάνει γι' αυτό. Λοιπόν, το βασικό μήνυμα είναι, είναι ότι πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, εποφελούμενοι από αυτή την χρονιά που δεν υπάρχουν εκλογές. Ευχαριστώ και είμαι πεπισμένο ότι όπω και τι προηγούμενε χρονίε θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τι άλλε πολιτικέ ομάδε για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρεντά. Λοιπόν, πριν να δώσουμε τον λόγο στους Κιώδης, ε, θα δώσουμε καταρχήν τον λόγο στον κύριο Πίτσουλο, που είναι πρόεδρος ε, της Επιτροπής Επιτροπής για τις σχέσεις με τη Βαυσίνη Σεγοβίνη. Ε, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Το σχέδιο έκθεσης ε, του κυρίου Πρέντα είναι πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις ε, για τη συμφωνία με την ε, Βοσνία Ριζεγοβίνη. Φυσικά, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν αμφιβολίες σε σχέση με τον ε, μελλοντική πορεία ε, της χώρας, αλλά θα πρέπει να ε, γίνουν οι μεταρρυθμίσεις από την κυβέρνηση. Θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία, να βελτιωθούν οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς... οι θετικές εξελίξεις σημαίνονται ταυτόχρονα με αρνητικά αποτελέσματα σε διάφορα πεδία και ε, είναι ανάμεκτα τα αισθήματα και στις γειτονικές χώρες της Βοσνίας Ζεγοβίνης σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις. Ε, πού χωλένει αυτός ο ευρωπαϊκός δρόμος της ε, Βοσνίας Ζεγοβίνης. ως βουλευτής και πρόεδρος αντιπροσωπείας για τη σχέση με τη Βοσνία Ζεγοβίνη μπορώ να σας πω ότι χρειάζεται ε, περαιτέρω προσπάθεια γιατί απέτυχε η προσπάθεια για μια κοινή ημερήσια διάταξη για ένα κοινό θεματολόγιο για τις επαφές μας. Έγιναν ε, διάφορες προσπάθειες για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς δεν καρποφόρησαν. Τα μέλη της αντιπροσωπείας από την Ρεπούμπλικα Σέρψκα μας ε, κατηγόρησαν ότι Υιοθετούμε μία ε, ε, πλημελή προσέγγιση όπως και σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε αντίστοιχες ε, διαδικασίες. Όμως υπάρχει ομοθυμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δεκτεί η σερβική πλευρά την πρότασή μας. Αλλιώς η αντιπροσωπεία δεν θα μπορέσει μέχρι νεοτέρας να συνεχίσει τις εργασίες της. Έχει Λοιπόν, διακοπεί η ε, διαδικασία. Σίγουρα δεν ε, μπορούμε και θα καταβάλουμε και κάθε προδυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να απεμπλακεί η κατάσταση, όμως σε μια, για μια μελλοντική λύση θα πρέπει να ξέρουμε, θα πρέπει να ρυθμιστούν πρώτα ζητήματα για το καλό των πολιτών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Σας ευχαριστούμε κύριο Παπαδάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο του εισηγητή είναι αρκετά ισορροπημένο και αγγίζει τα πιο σημαντικά ζητήματα που καλούμαστε να εξετάσουμε σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βοσνία. Θεωρώ ωστόσο πως σε ορισμένα σημεία οι σχετικές διατυπώσεις είναι τηλεγραφικές και ότι χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία και θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες. Καταρχήν πρέπει να αναδείξουμε περισσότερο ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας θα αλλάξει τα μέχρι σήμερα δεδομένα, θα επηρεάσει θετικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί πολιτεύονται στο εσωτερικό της χώρας και θα δώσει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον σε όλους τους πολίτες της χώρας ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους και την εθνική τους προέλευση. Διαπιστώσαμε ότι η παρουσίαση της αίτησης ένταξης επιτάχυνε τις συστημικά και πολιτικά δυσκολίες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και είχαμε επιτέλους μία λύση στο ζήτημα της προσαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης με τη Βοσνία Ζεγοβίνη το μηχανισμό για το συντονισμό και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της απογραφής του 2013. Επίσης, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στο κύριο κείμενο μία παράγραφος που να καλωσορίζει την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και που να εξετάζει και το ζήτημα της επικύρωσης. Πρέπει να υπάρξει μία αναφορά στην ανάγκη υιοθέτηση ενός στρατηγικού προγράμματος, σχεδίου, για τη σταδιακή ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό γεχτημένο, μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ των διάφορων Υπουργείων και συνιστοσών, γεγονός που τονίζει και η Επιτροπή στην έκθεσή της. Σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει για την εμπλοκή τους στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης και περαιτέρω ενταξιακή διαδικασίας. Σε σχέση με τις κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσέγγισης με μεγαλύτερη έφαση όμως στο κοινωνικό σκέλος. Σε ό,τι αφορά τις συνιστώσεις, καλωσορίζω την ισορροπημένη προσέγγιση του εισηγητή στη σχετική παράγραφο για το δημοψήφισμα στη Ρεπούμπλικα Σέρψκα, το οποίο βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν επικροτούμε αλλά το καταδικάζουμε εφόσον αποσκοπεί στην υπονόμευση της ενότητας της χώρας. Επιβάλλεται ωστόσο ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια προσέγγισης της Ρεπούμπλικα Σέρψκα και εμπλοκής στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις εθνικιστικές εξάρσεις και να σκεφτούν τον κοινόφιλο των πολιτών και οι γειτονικέ χώρε πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό. Βεβαίω, όμω, πολύ σωστά σημειώνει η εισηγητή, οι δυσκολίε παραμένουν και χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά και έμπρακτη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Αυτά προ τον παράγοντα δική μα πλευρά και ευχαριστώ τον εισηγητή που προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Κρίστιαν Πρέτα και τη Γραμματεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την έκθεση για την πρόοδο της Βοσνίας Ζεγοβίνης για το 2016. Εξ ονόματο ε, του ΕΛΚΕ θα θέλαμε να συγχαρούμε τη χώρα για την πρόοδο που σημειώθηκε το 2016. Υπολείπεται όμω πολύ δύσκολο έργο, είναι περίπλοκη η διαδικασία, λεπτά τα ζητήματα και δεν μας ξαφνιάζει το ότι δεν είναι επαρκής ε, η πρόοδο που έχει σημειωθεί για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο για την οικονομία, την καταπολέμηση οργανωμένης εγκληματικότητας, την αντιμετώπιση της διαφθόρας. Θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειε να βελτιωθεί ο συντονισμό ανάμεσα στι συναρμόδιε αρχές και μόνο βελτιώνοντα τη συνεργασία ανάμεσα στι διάφορε κοινότητε, θα μπορέσει να χαράξει την ε, πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η Βοσνία Ζεγοβίνη ενοποιήθηκε η διδακτέα ύλη σε ολόκληρη τη χώρα και αυτό το επικροτούμε. Έτσι, οι διάφορες κοινότητες ε, θα πρέπει να προσέξουν τι θα κάνουν με τις μειονότητες για να μην προκύψουν συγκρούσεις, να μην αποκλειστούν οι γλώσσες που μιλούν οι μειονότητες. Ε, είναι πάρα πολύ περίπλοκη διαδικασία και θα πρέπει στο ψήφισμα μας να συνυπολογίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο κύριο Βάγκουλ, ο οποίο θα πάρει το λόγο αντί για τον κύριο ράντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ζητά συγγνώμη ο κύριος Δράτος, ο σκιώδης ε, των φιλελευθέρων που δεν ήρθε. Εξ ονόματός του θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για την ακριβή και περιεκτική έκθεση που κατέθεσε. Ε, υποστηρίζουμε στεναρά το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας και υποστηρίζουμε και την πολιτική διεύρυνση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βοσνία Ζεγοβίνη έχει σημειώσει πρόοδο, όμω μην ξεχνάμε ότι οικονομικά και πολιτικά επικρατεί μεγάλη αστάθεια στη χώρα. Η Συμφωνία για το Μηχανισμό Συντονισμού θα έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος για τη διαδικασία κύρωση της συμφωνία ε, σύνδεση ε, και σταθεροποίηση. Ε, σε υψηλό επίπεδο δυσλειτουργεί η χώρα, πλήττεται από τη φτώχεια και οι δομέ δεν λειτουργούν. Δυστυχώς ε, συνεχίζουν εσωτερικές συγκρούσει και αυτές είναι πολύ μεγάλες προκλήσεις ε, κατά την πορεία της χώρας προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και σε άλλες χώρες, δύσκολα θα επιληθούν αυτές οι δυσκολίες Χρειάζεται επικοδομητικός διάλογος και συνεργασία ούτως ώστε να είναι μελλοντοστραφής η πολιτική και όχι στραμμένη προς το παρελθόν. Τους καλούμε να, ε, ε, κρίνουν, να υιοθετήσουν ε, τους κανόνες της Επιτροπής για την κύρωση της Συμφωνίας Σύνθεσης και Σταθεροποίησης. Εξακολουθεί να είναι ανεσυγητική η κατάσταση των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπιστέντων και η κατάσταση των εξαφανιστέντων. Ε, είναι πολύ αργή η δικαστική διαδικασία και οι αρχές θα πρέπει να πιέσουν τόσο ώστε να αντιδικοποιηθεί η συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες οντότητες. Θα ήθελα ίσως να προσθέσω από πλευρά μου και μία σκέψη θα βοηθήσει πάρα πολύ αν όλες οι εκθέσεις πρόοδοι για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να εμπεριέχουν μία σαφή θέση πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει για να ε, υπερβούν αυτές οι χώρες την τρέχουσα ε, προσφυγική κρίση. Ε, χωρίς να κάνουμε τους προφήτες, δεν είναι δύσκολο να προβλέψουμε ότι δεν θα επιληθεί σύντομα η κρίση. Για τα επόμενα χρόνια σίγουρα θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Ευχαριστούμε. Κύριε Σόλτες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα, τον εισηγητή, που προτίμασε αυτό το σχέδιο κειμένου. Πιστεύω ότι η έκθεση είναι πολύ σαφής, πολύ καλή και καλά ισορροπημένη. Υπογραμμίζει τις κύριες πτυχές που πρέπει η χώρα να βελτιώσει για να οδεύσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές το κείμενο. Και δεν ασκεί πιέση στη χώρα που αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Όταν συντάσσονται τέτοιες εκθέσεις είναι σημαντικό να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Η προσέγγιση που ακολουθείται από τον εισηγητή είναι ιδιαίτερα θετική και την υποστηρίζω πλήρω. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε την αρχή της ενότητας όπως είπαν και οι συνάδελφοι, πρέπει να γίνουν περισσότερα στο δημόσιο τομέα, στη δημόσια διοίκηση. και να διασφαλίσουμε το κράτος δικαίου. Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, όμως πολλά παραμένουν ακόμη να γίνουν. Και αυτός ο κατακαιρματισμός θα πρέπει κάπως ε, να διορθωθεί. Δεν έχουν εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις σε ορισμένου τομεί, επειδή είναι ιδιαίτερα κατακαιρματισμένη η χώρα. Ενίοτε αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται επαρκώς. Θέλω να τονίσω και κάτι ακόμη που δημιουργεί εμπόδια για την πρόοδο της χώρας, το οργανωμένο εγκλήμα και τη ευθορά. Αυτοί οι δύο τομείς είναι ένα μεγάλο εμπόδιο και σχετίζονται με τα δημοσιονομικά και την οικονομία. Έχουμε πολλές ε, υποθέσεις διαφθοράς που σχετίζονται με τη φοροδιαφυγή, τη φοροποφυγή κτλ. Γι' αυτό το λόγο η χώρα θα πρέπει να έχει μια κοινή προσέγγιση για να επιλύσει τα ζητήματα αυτά και θα πρέπει να επιλύσει και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το διορισμό δικαστών. Είδαμε ότι υπήρχαν προβλήματα στα δικαστήρια και στο δικαστικό σώμα και χωρίς τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος δεν θα σημειωθεί η πρόοδος αλλού. Πολλοί νέοι έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν τη χώρα και η Βοσνία Ερτσακοβίνη αντιμετωπίζει φυγή κεφάλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχε πολλή δουλειά να κάνει, γιατί οι νέοι είναι αυτοί που θα αλλάξουν τη χώρα και την πολιτική δομή της χώρας. Κάτι που έχει βελτιωθεί είναι το θέμα της απασχόλησης. Το ποσοστό της ανεργίας έχει μειωθεί το τελευταίο έτος, όμως και πάλι θα ήθελα να αναφέρεται στην έκθεση το περιβάλλον. Θα πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά στην έκθεση σχετικά με το περιβάλλον. Για αυτό θα προετοιμάσω κάποιες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως σε ό,τι αφορά τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, μάλιστα. Έχουμε και άλλους βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Κούκαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για ένα πολύ καλό πρώτο σχέδιο της έκθεσης. Νομίζω ότι ορθώς θίγει όλα τα σημαντικά ζητήματα και είναι και πολύ καλογραμμένο το κείμενο. Νωρίτερα φέτος η Βαρνία στην έκανε την αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έγινε δεκτή από το Συμβούλιο και κατόπιν της προσχώρησης ε, της Κροατρίας υπήρχε μια συμφωνία για, το, τη Συμφωνία Συνεργασίας και, το πρόγραμμα, για το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι σημαντικά βήματα προκειμένου να ανοιχτεί η διαδικασία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 μέχρι τώρα. Είναι ένα καλό έτος για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αληθεύει ότι υπήρχαν το Σεπτέμβριο κάποια προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη το δημοψήμισμα και ο εορτασμός της ε, Εθνικής Γιορτής ε, στην Ρεπούμπλικα Σέρσκα. Τώρα πρέπει να δούμε προς τα μπρος και να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά. Όλη η πολιτική ηγέτες θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπέθειες ε, για να εφαρμόσουν την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Χαίρομαι που σιγά σιγά αυξάνεται η ευθυγράμμιση της Βενής Αζεκοβίνης με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα η χώρα να παίξει ένα σημαντικό και επικοδομητικό ρόλο στα περιφερειακά ζητήματα. Υποστηρίζω πλήρως όσο είπε ο κύριος Πίτσουλα για τους διαδικούς κανόνες ε, του SCPC. Χωρίς να υιοθετηθεί αυτό, έχω κάποιες αμφιβολίες για το αν είναι νόμιμες οι δραστηριότητες της αντιπροσωπείας. Χάνουν την πολιτική του σημασία. Έτσι λοιπόν θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες και αυτό είναι μια υπόσχεση, όχι απειλή προς τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Πρέντα και όλους τους υπολείπους που, συμμετέχουν στην προετοιμασία της έκθεσης. Χαίρομαι που είμαστε τώρα πιο αισιόδοξοι όταν μιλάμε για τη Βοσνία ζεγοβίνη και ελπίζω ότι θα είμαστε και αισιόδοξοι και του χρόνου. Ένα έτος όπου δεν θα έχουμε εκλογές. Νομίζω ότι ο λαός αυτής της χώρας αξίζει περισσότερα και εμείς ε, θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για τη χώρα. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στις αρχές της χώρας να εργαστούν για το λαό τους, για τα έθνη τους. Θα πρέπει να κάνουν περισσότερα σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να δράξουν αυτή την ευκαιρία και να κάνουν περισσότερα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η διαφθορά αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για τη χώρα. Θα πρέπει να κάνουν περισσότερο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και να διασφαλίσουν ότι τα μέσα ενημέρωσης παραμένουν ελεύθερα. Πολλά πρέπει να γίνουν σε αυτό το τομέα, καθώς έχουν γίνει πολλά βήματα προς τα πίσω. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι η Επιτροπή προσχώρησης και σταθεροποίησης θα πρέπει να συσταθεί, θα πρέπει να συνομιλήσουμε με τους πολιτικούς στη χώρα και αυτό αποτελεί σίγουρα ένα μέσο που θα τους βοηθήσει. Γι' αυτό ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να απευθύνω έκκληση στους πολιτικούς να σταματήσουν ε, να εφαρμόζουν εθνικιστικές πολιτικές. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερος εθνικισμός στη χώρα. Και όπως ακούσαμε, οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, αν οι νέοι δεν έχουν πλέον όραμα για τη χώρα τους, τότε το μέλλον της χώρας θα τεθεί σε κίνδυνο. Και κάτι ακόμα, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών επίσης έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει πέρα από την κυβέρνηση. Και ελπίζω ότι και οι προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών θα ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν στην ε, κοινωνία της χώρας τους. Θα πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι και να εργαστούμε προς ένα πιο λαμπρό μέλλον για τη χώρα. Η Βοσνία Ριζεγοβίνη πρέπει να δώσει καλέ απαντήσει στο ρυθμολόγιο και αυτή είναι η οδό προ τα μπρο. Παρακαλώ, συνάδελφο Τσαφκά. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο Πρέντα για τις ε, ε, προσπάθειες, για τη δουλειά που έκανε. Η πορεία της Βοσνίας Ριζεγοβίνης προς το ΝΑΤΟ είναι σαφής. Αλλά παρά τις θετικές εξελίξεις στη χώρα πρέπει να τονίσουμε ότι εξεκολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις. Παρά τις ε, προόδους που σημειώθηκαν το 2014 και το 2015, η έκθεση προόδου δεν τονίζει ότι ε, ορισμένες ελλείψεις είναι συστημικές. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως είχε αναγνωρίσει το Κοινοβούλιο, ότι πρέπει να γίνουν εκβάθρον ε, μεταρρυθμίσεις μεταρρυθμίσει ορισμένου τομεί ε, για να επιτύχουμε το κράτος δικαίου. Και βεβαίως οι εσωτερικές διχόνοιες και πολιτικές διαφορές ε, παρεμποδίζουν αυτή την προσπάθεια. Και ο εκλογικός νόμος επίσης πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεκριμένος για τις τοπικές εκλογές, για τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Για πρώτη φορά από το 2004 στο Μόσταρα δεν, ήταν, δεν υπήρξε δυνατό να διεξαχθούν οι εκλογέ. Πρέπει να σταλεί σαφές πολιτικό μήνυμα προς την ε, Βοσνία Ζεγοβίνη. Επιπλέον, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη έναντι τη πολιτική εξουσία για να μπορεί να ε, επιτελεί το έργο τη. Και δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να ασχολείται με τη φυλάκιση ε, Κροατών σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν αποφασιστικά περισσότερες μεταρρυθμίσεις και να γίνουν και οι διαδικασίες ε, συμφιλίωσης. Λοιπόν, αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση. Τώρα έχουμε εδώ την κυρία Ματουέλα που θα ήθελα να της δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Πρέντα, για την ε, πολύ υψηλή επίπεδου και πολύ αντικειμενική έκθεσή του και ψήφισμα για την έκθεση 2016 για τη Βοσνία Ζεγοβένη. Το κείμενο είναι απόλυτα σύμφωνο με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της οποίας η έκθεση από τη μία συνεχάρει τη χώρα για τα θετικά που έχει επιτύχει και τόνισε και τα περαιτέρω βήματα που πρέπει ακόμη να γίνουν. Στο παρελθόν, τον παρελθόντα χρόνο δηλαδή, είδαμε ότι υπάρχει μια νέα δυναμική στη χώρα, διότι υπήρξαν ε, βασικές μεταρρυθμίσεις με βάση το θεματολόγιο. Έχουμε λοιπόν την εφαρμογή της, ε, του θεματολογίου μεταρρυθμίσεων που σε γενικέ γραμμές πάει καλά σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε το μηχανισμό συντονισμού που ήδη αναφέρθηκε ότι είναι ουσιώδης για να προχωρήσει η χώρα και έγινε μονογραφή του πρωτόκολλου ε, προσαρμογής ε, του Συμφώνου Σταθεροποίησης και ε, Εταιρικής Σχέσης. Και γι' αυτό το Συμβούλιο κάλεσε την Κομισιόν να υποβάλει γνώμη. Και ο Επίτροπος Χάν θα παρουσιάσει τα ερωτηματολόγια, το κατάλογο αρχικών ερωτημάτων την επόμενη εβδομάδα. Στις 9 Δεκεμβρίου θα την κοινοποιήσει στην Βυσνία, στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτό έχει τεράστια συμβολική σημασία, αλλά σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσει πολύ σιώδη δουλειά για όλε τι φάσει των κριτηρίων τη Κοπενχάγη. Και πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για να αντιμετωπιστούν τα βαθιά διαφορετικά προβλήματα που καθυστερούν την ε, πορεία της χώρας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κοινωνικο οικονομικέ προκλήσεις, το κράτος δικαίου και την μεταρρύθμιση της δημόσιας δίκησης. Ουσιώδες είναι να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης είναι προτεραιότητα. Και γιατί η χώρα φυσικά πρέπει να συνεργαστεί ενεργά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη φάση προετοιμασίας της ε, γνώμης. Και η ίδια η διαδικασία ε, εκπόνησης της γνώμης θα είναι ένα τεστ για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Και λίγο, επαναλαμβάνοντας, ότι δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει με τις σωστές συμβουλές, την τεχνική βοήθεια και την οικονομική βοήθεια η Κομισιόν λοιπόν τη Βοσνία Ζεγοβίνη για να επιτύχει τους στόχους της και ε, προς αυτή την κατεύθυνση το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει την πολύτιμη συνεργασία του. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που επέδειξαν ενδιαφέρον για τη Βοσνία Ζεγοβίνη και έκαναν πολύ ενδιαφέρουσες ε, και σημαντικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους που είπαν ότι ε, χρειάζονται συμπληρώσεις στο κείμενό μου. Φυσικά, μέσω τροπολογιών θα το συμπληρώσουμε. Χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες ε, επιλογές. είχαμε ε, με πολύ γενοδορία από ε, του αριθμού γραμμάτων που μπορούσε να περιέχει η εκθεσή μου, αλλά δεν μπορούσαμε να τα περιλάβουμε όλα και ελπίζω μέσω των τροπολογιών να συμπληρώσουμε αυτά που λείπουν. Σας ευχαριστώ για όλες τις προτάσεις που ήδη κάνατε κατά τη συζήτηση. Είμαι πεπισμένος ότι οι τροπολογίες θα διευκρινίσουν το κείμενο. Δεύτερον, Όταν ξεκίνησε η νέα πρωτοβουλία τη Βοσνία Ζεγοβίνη, υπενθυμίζω ότι ήταν πριν από δύο χρόνια, το 2014, στόχος μας ήταν να τους ζητήσουμε να κάνουν λιγότερα στην αρχή για να κάνουν περισσότερα μετά. Γι' αυτό είπα ότι αρχικά πρέπει να ασχοληθούμε με τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα και ας αφήσουμε για αργότερα τις μεταρρυθμίσεις και ιδιαίτερα τις συνταγματικές που είναι πάντα πιο περίπλοκες, πιο ευαίσθητες και που είναι πιο δύσκολο να τις ε, εφαρμόσουν οι πολιτικοί. Θεωρώ ότι αυτά που έγιναν είναι σημαντικά, αλλά απέχουμε πολύ ακόμη από ουσιώδεις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να εμείνουμε στην πορεία αυτή, να τους ανθαρρύνουμε να εμείνουν και εκείνοι και μόνο αργότερα Μπορούμε να ελπίζουμε ότι με μια πιο έντονη προσπάθεια η χώρα θα μπορέσει να αποφασίσει συνενετικά μεταρρυθμίσεις ιδιαίτερα συνταγματικές. Βεβαίως το θέμα είναι υποσυζήτηση αλλά τουλάχιστον δύο από τα κόμματα αρνούνται κατηγορηματικά κάθε συνταγματική μεταρρύθμιση. να τους προσφέρουμε εμείς λοιπόν ε, από τις Βρυξέλλες μια ευκαιρία για να μπλοκάρουν τις κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί βεβαίως ε, αν ξεκινήσουμε συζήτηση για συνταγματικές μεταρρυθμίσεις να μπλοκάρει όλα τα πάντα δεν νομίζω ότι είναι σωστή λύση. Το ερωτηματολόγιο που σε λίγο θα αποσταλεί θα περιέχει πάνω από 3.000 3.000 ερωτήσεις. Πολλές. Και εγώ, ε, ξέρετε, με κάθε μέτριο ε, μπορώ να τους δώσω μια συμβουλή. Ε, μπορούμε να ε, βασιστούμε στο ερωτηματολόγιο για την Ισλανδία. Η Ισλανδία ήταν χώρα υποψήφια και είχε απαντήσει με υποδειγματικό τρόπο το ερωτηματολόγιο. Ε, και ζητώ από τις αρχές να δουν την εμπειρία από τις χώρες γύρω, του, γύρω τους, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Ουγγαρία, αλλά γιατί να μην αξιοποιήσουν και το παράδειγμα των Ισλανδών που με θαυμάσιο τρόπο έκαναν ακριβώς αυτό που τους ζητήθηκε με ομάδες ε, ολιγάριθμες. Οι συνάδελφοι που εργάζονταν τότε μαζί με μένα για την Ισλανδία νομίζω συμφωνούν οι πολιτικοί και οι υπάλληλοι, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης στο Σαράγεφο θα μπορούσαν να αποφεληθούν από το αξιέπαινο παράδειγμα της Ισλανδίας όσον αφορά τη σοβαρότητα, το βάθος των απαντήσεων. Να μην σπαταλούν τον χρόνο τους σε μικροδιαφωνίες προσπαθώντας ο καθένας να διαφυλάξει το μαγαζάκι του. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε και λίγο ευρύτερα. Όχι μόνο γύρω μας ή στη διπλανή αυλή. Πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να έχουμε πιο ανοιχτή, πιο χαλαρή προσέγγιση. Είναι κάτι που και διανοητικά είναι πολύ θετικό για την πολιτική. Και θα συνεχίσω να τους συστήνω μια τέτοια προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη με αυτή την παθιασμένη απάντηση του κυρίου Πρέντα. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία είναι στις 10 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα για τις τροπολογίες. Και ολοκληρώσαμε εδώ αυτό το ζήτημα. Έχουμε τώρα την έκθεση που αφορά την Αλβανία εισηγητής είναι ο κύριος ε, Φλεκενστάιν. Πρόκειται για μια πρώτη συζήτηση και χωρίς να χάσουμε χρόνο θα του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να καλωσορίσω μια ομάδα νέων από την Αλβανία ε, με τίτλο EU Policy Hub, ε, κέντρο ενωσιακής πολιτικής έχουν σπουδάσει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέστρεψαν στη χώρα τους, όπου θέλουν να βοηθήσουν την ε, αναδιοργάνωση της χώρας. Αυτό είναι πολύ πιο ενθαρρυντικό μήνυμα, πολύ πιο ενθαρρυντικό από αυτά που μπορούμε να στείλουμε εμείς ως πολιτικοί, όταν οι νέοι μετά τις σπουδές τους γυρνάνε στη χώρα τους για να βοηθήσουν την βελτίωση της χώρας τους. Καλώς ήρθατε. Δεύτερον. Υπάρχουν πάντα αρκετές κρίσεις στα Βαλκάνια. Μία θα λήξει στις 11 Δεκεμβρίου στη Μακεδονία, λέει ο μιλητής. Στην Αλβανία γίνονται πολλές προόδοι όσον αφορά την εφαρμογή κάποιων βασικών προτεραιοτήτων. Τον περασμένο Ιούλιο αποφασίστηκε ομόφωνα η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και επίσης οι αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές από το Αλβανικό Κοινοβούλιο. Ομόφωνα, όπως είπα, με την σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων και της αντιπολίτευσης. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι νόμοι πέρασαν από τον έλεγχο των εισαγγελιών και έχουν εγκριθεί και διάφοροι εφαρμοστικοί νόμοι από το Κοινοβούλιο. Ορισμένοι ε, βουλευτές έθεσαν ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου κάποια θέματα τον Οκτώβριο, το οποίο τώρα αναμένει μια γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θεωρώ ότι παρά το ότι πολλά ακόμη δεν έχουν διορθωθεί και επί των οποίων θα αναφερθώ στην έκθεσή μου, θα έπρεπε να ξεκινήσουν ε, τάχιστα, όσο δυνατόν ταχύτερα, οι διαπραγματευτικές, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Εφόσον, βεβαίως, προχωρήσει στην πράξη η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Και εκεί ανήκει και αυτή η διαδικασία vetting, δηλαδή ελέγχου. Πρόκειται για σαφές μήνυμα ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή των διαπραγματεύσεων. Οπότε μπορούμε να συστήσουμε προς το Συμβούλιο, να συστήσει την Κομισιόν, να ξεκινήσει διαπραγματεύσει αν εφαρμοστούν αυτές οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και όχι να περιμένουμε το 18 όταν θα έχουμε την επόμενη έκθεση. Το θέμα είναι και για μας να παραμείνουμε αξιόπιστοι. Ήταν δύσκολη απόφαση αυτή που έλαβε το Κοινοβούλιο ιδιαίτερα για την αντιπολίτευση, που συμφώνησε σε όλα. Και του είπαμε, α, αυτή είναι η ορθή και θα το αναγνωρίσουμε. Θα αναγνωρίσουμε τι προσπάθειές σα. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν τώρα να θέσουμε επιπλέον προποθέσει, Δεν θα ήταν δίκαιο. Παρ' όλα αυτά είναι σαφέ ότι χρειάζονται επιγόντω και περαιτέρω διαπραγματεύσει και περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να καταπολεμηθεί η διαφθορά ή το οργανωμένο έγκλημα. Και ο εκλογικό νόμο επίση πρέπει να εφαρμοστεί γιατί περιμένουμε του χρόνου να γίνουν ελεύθερες εκλογές χωρίς αγορά ψήφων και άλλα τέτοια φαινόμενα ανοθείας που έχουν ε, σημειωθεί στο παρελθόν. Είναι θέμα δικαιωμάτων μειονοτήτων που βεβαίως πρέπει να γίνονται σεβαστά και να αντιμετωπιστεί και η εγκληματικότητα. Να καταλήξουμε με δύο θετικά. Πρώτον, η Αλβανία έχει ένα σταθερό και σταθεροποιητικό ρόλο μαζί με την Σερβία για να υπάρξει συμφιλίωση στην περιοχή και τελευταία ο ρόλος αυτός έχει ενισχυθεί. Η περιφερειακή ανταλλαγή νέων. Υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα στα Τύρανα. Είναι παράδειγμα αυτό και το θεωρούμε πολύ σημαντικό διότι όταν οι νέοι δεν ε, ε, γνωρίζουν ένα τον άλλον, δεν είναι δυνατόν να ε, ξεπεραστούν οι παλιές ε, προκαταλήψεις. Η Αλβανία είναι όχι μόνο για τις Βρυξέλλες, αλλά και για την Ουάσιγκτον ένας αξιόπιστος εταίρος. Χαίρομαι για την πολύ καλή συνεργασία με τους σκιώδεις συζητητές ως συνήθως. Ίσως να μην περιέχονται όλα όσα θα ήθελα στην έκθεσή μου, γιατί έπρεπε να έχει συγκεκριμένο μήκος, αλλά είμαι σίγουρος ότι επίσης μέσω των τροπολογιών και από άλλα κόμματα πολλά σημεία θα προσταθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μακνούτ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους κοιόδης εισηγητές που είναι εδώ. Καταρχήν, κύριο Κούπερ. Ευχαριστώ Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, πρώτα απ' όλα. Έκανε σημαντικές προσπάθειες ε, για να προετοιμάσει αυτή την ε, ακριβή και ισορροπή έκθεση για την Αλβανία. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το σταθεροποιητικό ρόλο της Αλβανίας στη περιοχή και την πλήρη ευθυγράμμισή της με τις δηλώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταδεικνύουν την προσήλωσή της ε, στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ε, ήταν πολύ θετική η πρόοδο σε σχέση με τα κριτήρια για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μετά από την έγκριση των πέντε βασικών προτεραιότητων και την έγκριση της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συστήσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με προσχώρηση της Αλβανίας και χαίρομαι που συμφωνεί ο κύριος Φλέκενστάιν, όπως αποτυπώνεται και στην έκθεσή του. Ήρθε η ώρα για να αρχίσει η διαδικασία αυτή στην Αλβανία. Φυσικά ε, πολλά πρέπει να γίνουν και οι βρεχόμενες προεδρικέ και βουλευτικέ εκλογέ το 2017 θα είναι η πραγματική λιδία λίθος για την ετοιμότητα τη χώρα ε, για την έναρξη των διαδικασιών προσχώρηση. Ελεύθερες ε, και δίκαιες εκλογές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την Αλβανία, ώστε να μπορέσει να προοδεύσει και θα πρέπει να το επισημάνουμε στην έκθεση. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ο επικοδομητικός διάλογος ανάμεσα ε, στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση έχουν κέρια σημασία, κυρίως μετά τη δήλωση της αντιπολίτευσης για την αποχή ε, στην εκλογική διαδικασία αν δεν πληρούνται δύο προϋποθέσεις η εφαρμογή της νομοθεσίας για την αποποινικοποίηση και η εγγύηση για των καθαρών ε, και δίκαιων διαφανών εκλογών πάνω από 2 εκατομμύρια Αλβανοί ομογενείς δεν μπορούν να ψηφίσουν ενώ είναι βασικό κατοχυρωμένο σταγματικό δικαίωμα και η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει τι απαιτούμενε μεταρρυθμίσεις ώστε να τους δώσει αυτή την ευκαιρία. Μόνο τότε θα είναι πλήρως δημοκρατικές οι εκλογές στην Αλβανία. Τέλος, υπάρχουν πολλές προκλήσεις ακόμη. Έχουν γίνει όμως βήματα από την κυβέρνηση για να αντιμετωπιστούν. Παραδείγματο χάρη, προσπάθεια για την αντιμετώπιση της Ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης, του βίου εξτρεμισμού και έγκριση βασικών νομοθετημάτων για την καταπολέμηση της ε, ε, διαφθοράς. Και ε, ε, την ενσωμάτωση στην κοινωνία όλων των μειονοτήτων. Ευχαριστούμε και προσβλέπουμε στην μελλοντική συνεργασία του κύριο κ. Φλέγκεσταν και τους λοιπούς σκιώδης. Ο κ. Χατζηγεωργίου. Uh, Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Σταϊνό με πολύ σημαντική δουλειά που έκανε. Ε, όμως θα χρειαστεί να θέσουμε κάποια ζητήματα για την Αλβανία. Θα πρέπει να ε, ε, συνεχίσει τη διαδικασία προσχώρησης ε, υλοποιώντας περαιτέρω μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζοντας την οργανωμένη εγκληματικότητα στη χώρα και βελτιώνοντας επιδόσεις τους για την ελευθερία έκφρασης. Επίσης, σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αυτό είναι ένα ε, σημείο κέρια σημασία για μας. Και χρειάζεται ε, επίσης κατάλληλη απόκριση. Τι έγινε με αυτή την κατεδάφιση 20 σπιτιών ε, των πολιτών της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες Και μπορούμε να πούμε ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με επικοδομητικό πνεύμα, ώστε να ε, έχει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον η Αλβανία. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στους βουλευτές που τον έχουν ζητήσει, ο κ. Σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο ε, σε τομείς όπως η δικαιοσύνη και η καταπολέμηση της ε, διαφθοράς όμως έχουμε και περιστατικά τα οποία αποδεικνύουν μια έξαρση του εθνικισμού, όπως είναι η σύλληψη δύο υπαλλήλων του Αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στην προσπάθειά τους να μεταφέρουν προπαγανδιστικό υλικό για τη Μεγάλη Αλβανία, ε, χάρτες ε, προκειμένου, ώστε αυτό να μοιραστεί στους μαθητές αλβανικής καταγωγής που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία. Αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο και σίγουρα δεν συμβαδίζει με την υποχρέωση για σχέσει καλή γειτονία. Γι' αυτό το λόγο θα καταθέσω και ανάλογε τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ τον εισηγητή και τη γραμματεία για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής από πλευράς ε, του ECR. Συγχαίρουμε την ε, Αλβανία για την πρόοδο που έχει κάνει. Και θέλουμε να ε, αναφέρουμε ότι είμαστε αλληλέγγυη με τον αλβανικό λαό η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, βήμα για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στην απονομή δικαιοσύνης ε, και η πρόταση που θα σημειωθεί ε, του χρόνου είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουν να αρχίσουν οι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση. Ε, θα πρέπει να αναλυθούν μέτρα για την προστασία των μειονοτήτων από την κυβέρνηση. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών για τη συγκρότηση ειδική επιτροπής για τις γλώσσες των μειονοτήτων έχουμε σε δύο περιοχές ε, ε, βουλγαρικές μειονότητες που δεν έχουν όμως αναγνωριστεί, δεν έχουν το αντίστοιχο ε, καθεστώς. Θα ήθελα πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση να ζητήσω μετεβιτάσεις από τις αρχές ε, να αναγνωρίσουν αυτές τις ε, πληθυσμιακές ομάδες ως μειονότητες. Κυρία Σακοράφη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φλανιεστάιν για τη δουλειά που έχει κάνει στο προσχέδιο. Ε, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, αν δεν χρειάζονται κιόλα ε, συμπλήρωση. Προσωπικά, δύο ζητήματα θα ήθελα να επισημάνω, που τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο έχει να κάνει με τον πλήρη σεβασμό των μειονοτήτων, όπω έχει ξανααναφερθεί προηγουμένω, και το δεύτερο με την ανάπτυξη και την διατήρηση των σχέσεων καλή γειτονία. Πρόκειται για δύο θεμελιώδη ενταξιακά κριτήρια που η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει από τις συνθήκες να τηρεί, να, τις, να τα διασφαλίζει, ότι στις σχέσεις με τρίτες χώρες, αλλά ιδιαίτερα κατά την ενταξιακή διαδικασία αυτά τα δύο κριτήρια θα γίνονται απόλυτα σεβαστά. Η Αλβανία, όπως είναι πολύ σωστά επισημάνεται και η Φλιγκεστάιν, θα πρέπει να εργαστεί όπως οφείλει για την βελτίωση των συνθήκων όλων των μειονοτήτων στη χώρα. Ενώ όμως αναφέρεστε σε Άλλε μειονότητε, παραδείγματο χάρη το, του Ρωμά, δεν αναφέρεται τίποτα για την ελληνική μειονότητα, όπω δεν αναφέρεται και τίποτα για την υποχρέωση τη χώρα να ενισχύσει όπω οφείλει το νομικό καθεστώ που διασφαλίζει την προστασία των μειονοτήτων και ιδιαίτερα την προστασία του δικαιώματό του στην ιδιοκτησία. Και θα αναφερθώ και εγώ στο θέμα των, ε, των 19 οικογενειών της ελληνικής μειονότητας, τα οποία η κυβέρνηση, στις οποίες η κυβέρνηση έδωσε προθεσμία πέντε ημερών για να εκενώσουν τις κατοικίες τους που προορίζονταν για κατεδάφιση, μια ενέργεια που συνιστά καταφανή παραβίαση των, διεθνών, των αναγνωρισμένων ε, δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Επιπλέον, υπάρχει παντελής έλλειψη... Επιπλέον, υπάρχει παντελή έλλειψη αναφορά στην πρόοδο σχέσεων καλή γειτονία και ιδιαίτερα στην ανάγκη αποφυγή πράξεων και δηλώσεων που επηρεάζουν αρνητικά τι σχέσει αυτέ. Και το λέω αυτό πιστεύοντα ότι είστε ενήμερο και δεν αναφερθήκατε σε αυτό, ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται έξαρση αλυτρωτικών αναφορών τόσο από τον Αλβανό Πρωθυπουργό, όσο και από αρκετά μέλη τη ε, κυβέρνησή του εναντίον τη Ελλάδα. Εγώ προσωπικά θα καταθέσω τι σχετικέ τροπολογίε, ακριβώ γιατί πιστεύω ότι τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να προτάσσονται πάντα για να μην αφήνεται κανένα περιθώριο να παίζονται μικροπολιτικά παιχνίδια από τι εκάστοτε κυβερνήσει των χωρών αυτών. Σα ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε, κύριε Σόλτε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να να εκφράσω μια σοβαρή ανησυχία σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, προστασίας της φύσης. Θα ήθελα να αναφέρω ότι 44 από το 71, 44 71 υδροελεκτρικά εργοστάσια κατασκευάζονται τώρα σε προστατευόμενες περιοχές και από τις ΜΚΟ λάβαμε πολλές επιστολές σε ό,τι αφορά τον ποταμό Βιώσα. Είναι ένας ε, σημαντικός ε, ποταμός στην Ευρώπη, είναι σκανδαλώδες αυτό και πρέπει να πούμε στην αλβανική κυβέρνηση να σταματήσει αυτά τα μη ελεγχόμενα έργα για την υδρολεκτική ενέργεια και να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτά δεν συνάδουν με το κεκτημένο. Ούτε με την ε, οδηγία της προστασίας της ε, φύσης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, θα πρέπει να σκεσπίσει για να γίνουν σεβαστά τα πρότυπά μας και τα διεθνή πρότυπα και θα ήθελα να αναφερθώ και στο ρόλο των ευρωπαϊκών τραπεζών σε αυτό το project που έχει συγκεκριμένο ρόλο. Επίσης, ο τοπικός πληθυσμός θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία Διαφορετικά θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση άγριας δύσης εκεί και θα πρέπει να δοθεί τέλος. Ο ποταμός στο οποίο αναφέρθηκε ο κυρίος είναι ο ΑΟΣ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής ανέφερε σημεία στα οποία υπάρχει πρόοδος στην προσπάθεια της Αλβανίας να ενταχθεί στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέφερε και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν επιπλέον. Δεν ανέφερε όμως ένα βασικό στοιχείο το οποίο έχει ε, να κάνει με την υποχρέωση της Αλβανίας να διατηρεί σχέσεις καλής γειτονίας με όλες τις γειτονικέ της χώρες. Θα αναφερθώ και εγώ στις ε, ε, στους χάρτες με την ε, Μεγάλη Αλβανία οι οποίοι κυκλοφορούν κατά καιρού και εκεί υπάρχουν εδάφη από όλες τις γειτονικές χώρες της Αλβανίας. Δηλαδή την Ελλάδα, τα Σκόπια και τη Σερβία. Με αυτή λοιπόν την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Αλβανίας κάθε άλλο παρά σταθεροποιητικό παράγοντα για την περιοχή των Βαλκανίων αποτελεί. Πρόσφατα επίσης ο Πρωθυπουργό της Αλβαγίας, χωρίς να υπάρχει λόγος, εξέφρασε επικρατικέ βλέψεις της χώρας του κατά της Ελλάδος και προσέβαλε την ιστορία της Ελλάδος αναφέροντας διάφορες ιστορικές ανακρίβειες. Εάν σε αυτά προσθέσουμε και την επαναχώρηση της Αλβανίας για να καθορίσει με την Ελλάδα την ΑΟΣ των δύο χωρών προκειμένου να ε, υποστηρίξει την τουρκική πολιτική επάνω σε αυτό το θέμα καθώς επίσης και την παραβίαση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Υπήρου αναφέρθηκαν οι καταδαφίσεις σπιτιών, έχουν καταδαφιστεί ναοί, δεν επιτρέπεται στους ε, ελληνική καταγωγή, αλφανούς υπηκούς να εγγράφονται στους ε, εκλογικούς καταλόγους, γίνονται ομές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των εκλογών στην εκλογική διαδικασία. Εάν λοιπόν όλα αυτά τα συνυπολογίσουμε, θα δούμε ότι η Αλβανία ακόμη δεν είναι έτοιμη για να αρχίσει τις ενταξιακές διαδικασίες. Και στο σημείο αυτό για να τελειώσω θα αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει με την Αλβανία το ίδιο λάθος το οποίο έκανε και με την Τουρκία. έχετε να παραβιάζει τις αρχές που πρέπει και υποχρεούται να εφαρμόζει προκειμένου να πληρεί τα κριτήρια της συνδίκης Κοπενχάγης με αποτέλεσμα να αποθρασύνει την Αλβανία. Πότε επιτέλους θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πείσει την αλβανική κυβέρνηση ότι είναι προς το δικό της συμφέρον να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία έχει ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αλβανία. Και έτσι όπως σωθούνται τα πράγματα υποχρεώνει την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να προβάλλει βέτο στις διαδικασίες εντάξεως. Αυτή θα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη αν τα πράγματα συνεχίσουν να κινούνται με αυτόν τον ρυθμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κύριε Θεοχάρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Φλίγκενστάιν για την έκθεση που μας έχει καταθέσει και να καλωρίσω και εγώ με τη σειρά μου τους Αλβανούς νέους οι οποίοι με ξεχωριστή μόρφωση αντιλαμβάνονται ότι το μέλλον της χώρας τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εργαστούν με ζήλο για να μπορέσει η χώρα τους να φτάσει στα ευρωπαϊκά επίπεδα που θα τις επιτρέψουν να γίνει ένα πλήρες και ισότιμο μέλος της ε, Ένωσης. Ωστόσο, είμαι υποχρεωμένη να υπερασπιστώ την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας για την οποία κανείς δεν μιλάει. Ασχολούμαστε με πολλές άλλες μειονότητες, αλλά όχι με την ελληνική Θέλω να σας πω ότι η ελληνική μειονότητα κινδυνεύει άμεσα. Το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο με τις μετακινήσεις Κωσοβάρων που δεν είναι καν Αλβανοί πολίτες προς τις νότιες περιοχές της ε, Αλβανίας καθώς επίσης και τη μετεγκατάσταση ένα καλασικό παράδειγμα των προσφύγων των Σιητών από το Ασράφ στα νότια των Τυράννων. Ε, δεν λέει κανείς να μην προστατευτούν πρόσφυγες, αλλά η πολιτική είναι να διοχετευτούν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες από το Ασράφ στις νότιες περιοχές της χώρας. Η διακρίση σε βάρος των Ελλήνων της Αλβανίας, οι οποίοι είναι και Ευρωπαίοι πολίτες, γιατί όταν η Αλβανία περνούσε την πιο μεγάλη οικονομική κρίση, όλος ο αλβανικός πληθυσμός, Έλληνες και Αλβανοί, είχαν μετακινηθεί στην Αθήνα και οι Αλβανοί έχουν ευεργετηθεί πάρα πολύ από το ελληνικό κράτος και συνεπώς είναι άδικα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε βάρος των Ελλήνων της Αλβανίας αλλά και σε βάρος της, ε, σε βάρος της Ελλάδας δεν μπορούν να, να μπουν στην διοικητική δομή της χώρας, δεν μπορούν να γίνουν στρατιωτικοί, δεν μπορούν να γίνουν δικαστές, δεν μπορούν να μπουν στο ε, στις διάφορες υπηρεσίες. Δεν μπορούν να γίνουν πανεπιστημιακοί. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ελληνικών σχολείων στην Αλβανία και σας το έχω αποδείξει και την προηγούμενη φορά. Πέρα από το γεγονό ότι η Αλβανία συνεχώ προβάλλει εδαφικέ διεκδικήσει σε βάρο τη Ελλάδα, έχει ε, αποσταθεροποιητική διείσδυση μέσα στα Σκόπια και ε, επέζει ένα πολύ επικίνδυνο ρόλο στο Κόσοβο. Δεν μπορώ να αγνοήσω και τον την τουρκική διοίκηση, την Ισλαμική διοίκηση μέσα, την Ισλαμική διείσδυση μέσα στην ε, Αλβανία με την ίδρυση των, αλβανικών, των ε, μουσουλμανικών σχολείων και νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι αν η Αλβανία δεν λάβει τα σωστά μέτρα, αυτά που αναφέρει ο κύριος Φίνγκεσταν για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, για την, ε, για την βελτίωση της διοίκησης και των νόμων για τον, ε, για εκλογικό νόμο. Ε, δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια θέση ε, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θέλω να τελειώσω λέγοντας σας ότι όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές συνηθίζουν να μετακινούν διοικητικά οικισμούς με αλβανικό πληθυσμό σε περιοχές που κλασικά ελέγχονταν από, τον ελληνικό, από τους Έλληνες αυτόχθονες κατοίκους για να μην μπορεί ποτέ να εκλεγεί δήμαρχος ή ε, πρόεδρος της κοινότητας μιας περιοχής ελληνικής καταγωγής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Ο Μαρίας, Μαριάς. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Pardon? Do I have the floor? Okay, okay. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ τον συνάλφο τον... Να συγχαρώ τον συνάλφο τον κύριο Φλέγκεστάιν για την έκθεσή του και να επισημάνω και εγώ αυτά που έχω πει αρκετές φορές στην Ολομέλεια για το θέμα της ε, Αλβανίας. Δεν είναι κάτι καινούριο που θα πω, το έχω πει στην Ολομέλεια, μερικές φορές ο συνάδελφος με έχει ακούσει, όπως και ο κύριος Πρέντα που είναι συχνά μέσα στην ε, Ολομέλεια. Υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο θέμα είναι η προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Υπήρου. Και εδώ έχουμε μια συνεχή παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων με αποκορύφωμα τα όσα συνέβησαν από το 2015 και μετά. Έχουμε την κατεδάφιση της Εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου στο χωριό Δρυμάδες, Έχουμε την αφαίρεση ιδιοκτησιών 123 τίτλων ιδιοκτησίας ελληνικών οικογενειών στο χωριό Δρυμάδες. Για το θέμα αυτό έκανα ερώτηση στις αρχές ε, Απριλίου και υπάρχει και απάντηση του κυρίου Χάν, ο οποίος επισημαίνει ότι η Αλβανία οφείλει να ε, σεβαστεί τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Επιπλέον έχουμε το τελευταίο φαινόμενο της απειλής για κατεδάφιση 19 κατοικιών ε, στην περιοχή του οικισμού σπηλαίων της Χιμάρας. Αυτό δείχνει ότι η κατάσταση δεν βαίνει καλώς όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Υπήρου. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ο εισηγητή θα πρέπει σοβαρά να το λάβει υπόψη, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Επομένως, σε αυτού του θέματος θέλουμε να υπάρχει ε, αναφορά. Θα καταθέσουμε βεβαίως και τροπολογίες, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει. Το δεύτερο θέμα που έχει σχέση πάλι με την ελληνική εθνική μειονότητα της Βόρειου είναι τα δικαιώματά της. Αν μπορεί στην πράξη να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα. Και έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα. Αντίθετα, ε, πάρα πολλοί οι κάτοικοι της Αλβανίας όταν ήρθαν στη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν, τα παιδιά τους να μορφωθούν, να αποκτήσουν χρήματα, να επενδύσουν αυτά τα χρήματα στην Αλβανία. Νομίζω λοιπόν ότι και ο αλβανικός λαός δεν επιτρέπει στην κυβέρνησή του αυτή την, την απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στην ελληνική εθνική μειονότητα της Βορείου Πύρου. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν, τις σχέσεις καλής γειτονίας. Πρώτη παρατήρηση, όπως είπε και ο κύριος Μπαν Κιμούν, η Αλβανία παρανόμως έκλεισε τα σύνορά της και δεν αφήνει τους πρόσφυγες να περάσουν δια της Βαλκανικής οδού. Και αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο και παράνομο. Δεύτερον, επιλεκτικά μεταφέρει όμως άλλους πρόσφυγες, ε, όπως ε, ανέφερε η συνάδελφος η κυρία Θεοχάρους. Τρίτον, μας ανησυχεί η αντίληψη περί μεγάλης Αλβανίας, που την έχουμε ακούσει αρκετές φορές, αλλά πλέον υπάρχει μια τεράστια έξαρση από πλευράς του κυρίου Ράμα, ο οποίος διατυπώνει ανιστόρητες απόψεις ακόμη και για την Ακρόπολη, διαμορφώνει ένα κλίμα ιστερίας ανθεληνικής ε, μέσα στην ίδια την ε, Αλβανία και επίσης ισχυρίζεται ε, διάφορα περί και για να εξηγήσω, αν δεν το έχετε ακούσει εδώ, οι Τσάμιδες ήταν συνεργάτες των SS ε, κατά τη διάρκεια της κατοχής του 1941-44 έδρασαν μαζί με τα SS και έφυγαν μαζί με τα SS προκειμένου να γλιτώσουν. Έχουν καταδικαστεί όμως από τα δικαστήρια της Ελλάδος ως συνεργάτες των SS και γι' αυτό είναι απίθανο τώρα αυτό που συμβαίνει, ο κύριος Ράμα να στηρίζει τους τσάμιδες και να στηρίζει τις δίθεν αξιώσεις τους. Αυτά λοιπόν είναι ξεκάθαρα πράγματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν και από την Επιτροπή μας και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν δεχόμαστε ούτε τις απειλές του κυρίου Ράμα, ούτε τις παράνομες διεκδικήσεις του. Αυτό λοιπόν το κλίμα δείχνει ότι δεν μπορεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις η Αλβανία να προχωρήσει στην ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο από όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντα κυρία Πουτουέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, προετοιμασία μιας ε, πολύ ισορροπημένης έκθεσης για την Αλβανία. Αυτό το σχέδιο έκθεσης συνοψίζει πολύ καλά τα πιο σημαντικά μηνύματα για την Αλβανία ουσιαστικά σχολιάζει την αποφασιστική πρόοδο του σχολείου και τονίζει τι ε, κύριε προτεραιότητε μεταρρυθμίσεων για την επόμενη περίοδο. Συνάδουν αυτά τα μηνύματα με αυτά τη Κομισιόν και επικεντρώνονται στην εφαρμογή τη ε, μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο, την καταπολέμηση τη διαφθορά και του οργανωμένου κλίματο, ε, την επιβολή των, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα θέματα όπως είναι η κλοκή μεταρρύθμιση και η εφαρμογή της διαδικασίας αποποινικοποίησης σημειώνοντας σταθερή πρόοδο από το 2014 που απέκτησε το καθεστώς ε, η Ελβενία έχει ε, παρουσιάσει αυτά αποτελέσματα και φυσικά τα πιο αξιοσημείωτα ήταν η υιοθέτηση των συνταγματικών ε, τροπολογιών και η συνολική μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος. Γι' αυτό το θέμα η Κομισιόν έχει ε, κάνει πρόσθετη σύσταση για να ανοίξουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, καθώς έχει σημειωθεί απτή πρόοδος ε, στην διαδικασία που αφορά την μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος και τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Αυτό ε, είναι απαραίτητο για την επιβολή του κράτους δικαίου στην Αλβανία και είναι σχετικό και για την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, συμφωνούμε για τον επικοδομητικό ρόλο που παίζει η Αλβανία στην περιοχή, καθώς και την δέσμευση ε, με την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Κομισιόν θεωρεί ότι υπάρχει επικοδομητικός διάλογος και θα είναι σημαντικός όχι μόνο για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων αυτών και για την όλη διαδικασία προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο πλαίσιο της διαδικασίας ε, της Επιτροπής, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Μπορούμε να δώσουμε χρήσιμη πολιτική καθοδήγηση για την ε, ευαίσθητη περίοδο που ακολουθεί και αναμένουμε να έχουμε μια καρποφόρο συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, είναι μια πρώτη συζήτηση αυτή και βεβαίως ε, θα πρέπει να συνεννοηθούμε και για τις τροπολογίες με βάση τις οποίες θα συζητήσουμε σε περισσότερο βάθος. Θα είμαι πολύ σύντομος. Κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, ε, ε, ίσως έγινε λάθος. Τα κριτήρια της Κοπεχάγης πρέπει να τηρούνται όταν κάποιος θέλει να μπει στην Ένωση, όχι όταν ξεκινούν διαπραγματεύσεις. Εδώ πρέπει να έγινε λάθος ε, αποφάσισαν μια τροποποίηση, μια μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη, την οποία άλλε χώρε αποφάσισαν όταν είχαν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσει. Γιατί λοιπόν να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σωστή σειρά. Πρώτο είναι η εκκίνηση των πραγματεύσεων και ό,τι πρέπει να τηρηθεί, πρέπει να τηρηθεί. Εάν στο τέλο πρέπει κανεί να γίνει μέλο τη Ένωση. Δεύτερον, ναι, ισχύει. Και το ανέφερα σύντομα και μπορούμε να το επεκτείνουμε μετά από ζητήσει. Βέβαια, όλα δεν, δεν πάνε καλά, όχι. Ορισμένα δεν είναι πραγματικά καθόλου καλά. Και καταλαβαίνω βέβαια γιατί συμβαίνουν ορισμένα πράγματα. Όταν για παράδειγμα καταταφίζονται αυθαίρετα, δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Να μπαίνει κάποιος ε, και να σου λέει ε, σήκω και φύγε και θα σου κρεμίσουμε το σπίτι ανεξάρτητα αν είναι αυθαίρετο οικοδομημένο από έναν ε, Έλληνα της Αλβανίας, από ένα μέλος της ελληνικής μειονότητας ή από άλλον. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται με τη σωστή νομική ασφάλεια. Πρέπει η διαδικασία να είναι κανονική. Αυτό είναι αναμφίβολο. Μια φράση για το τέλος. Βεβαίως ε, είδα ότι πολλοί Έλληνες συνάδελφοι πήραν το λόγο. Αυτό το βλέπουμε και για άλλα θέματα. Κανένα κράτος μέλος δεν ε, αισθάνεται να πιέζεται τόσο πολύ από άλλους όσο οι Έλληνες συνάδελφοι. Αυτό ισχύει για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ισχύει για την Αλβανία, ισχύει για την Τουρκία και πολύ συχνά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν πολλά ανεπίλητα θέματα με τη δική σας μειονότητα, ε, κυρίως στα Βαλκάνια. Γι' αυτό προτείνω και δεν θέλω να το ε, εκλάβετε ηρωνικά ή ίσως επίκριση. Εμείς ε, θα πρέπει ίσως στο διευρυμένο προεδρείο μας να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε ειδικά με τους Έλληνες συναδέλφους να συζητήσουμε τα προβλήματα που βλέπουν οι Έλληνες στην Αλβανία, τη Μακεδονία αλλιομιλητής και αλλού. Γιατί νομίζω ότι καθήκον μας είναι να λύνουμε και τα διμερεί προβλήματα και να λαμβάνουμε σαφή θέση, ούτω ώστε συνολικά η διαδικασία να κολλάει πάντα στο ίδιο σημείο. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε συγκεκριμένα αυτό, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ούτω ώστε να τα συζητήσουμε μεταξύ μας περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Και θα το συζητήσω με τον κύριο Μπροκ και το Προεδρείο και θα τους κάνω κάποιες προτάσεις. Ευχαριστώ Κνούτ να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία είναι στις 10 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι για την κατάθεση τροπολογιών. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και τη συζήτηση για την Ελβανία. Έχουμε ένα τελευταίο σημείο στην ημερησία διάταξη, Αντιλογή απόψεων σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Μολδαβία. Όπως ε, ξέρετε, κέρδισε ο Γκορτοντών με το 52,16% ψήφων. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σόλτες για μια σχετική ενημέρωση. Και κατόπιν ε, θα πάρει το λόγο ποιος το επιθυμεί. Έχουμε 14 λεπτά στη διάθεσή μας ε, το πολύ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 6. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να μιλήσω για την ε, αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρατηρήσουμε το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Μολδαβία που έλαβαν χώρα στις 13 Νοεμβρίου. Τα μέλη της ε, Διεθνούς Αποστολής Εκλογικής Παρατηρήσης συνάντησαν και τους διποψηφίους Ιγκορντοντών και Μαϊα Σάντου. Μία μέρα πριν από τις εκλογές, ο Ιγκορντοντών εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα κέρδιζε τις εκλογές ε, με 800.000 ε, ε, ψήφους, έναν εκατομμύριο ψήφους και ξέρουμε ότι υπήρχε μικρό περιθώριο μεταξύ των δύο. Επίσης αναφέρθηκαν κάποιες καταγγελίες ότι κάποιοι φοιτητές δεν μπορούσαν να ψηφίσουν. Επίσης ένιωθε ότι υπήρξε εισαγωγή διάκρισης ε, στο γεγονός ότι σε 92 ε, ε, εκλογικά κέντρα είχαν ανοίξει δική χώρα και μόνο 18 στη Ρωσία. Επίσης θεωρήθηκε ότι είχε περάσει, είχαν περάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωση σε πάρα πολλέ γραμμές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκστρατείας. Απ' την άλλη η Μάγια Σάντου τόνισε ε, ότι ήταν ε, διαφανής η εκλογική της εκστρατεία και ότι χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, για να κινητοποιήσει την υποστήριξη, όμως είπε ότι ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσει την εκστρατεία του αντιπάλου της και μάλιστα και τις δηλώσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας εναντίον της. Ε, δηλώσεις κατά της Μάγια Σάντου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συμπεριλάμβαναν και μία ε, συμφωνία ε, με την κυρία Μέρκελ να μεταφερθούν πρόσφυγες στη Μολδαβία και την ρώτησαν για το πόσο είναι κατάλληλη να αναλάβει τέτοια καθήκοντα καθώς ήταν ανήπαντρη και χωρίς παιδιά. Οι διεθνείς παρατηρητές παρατήρησαν την αρνητική τακτική που χρησιμοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε σεξιστική γλώσσα και κάποια στερεότυπα κατά του φίλου και κάποιες προσβλητικές δηλώσεις. Ο κύριος Ντοντών από το Σοσιαλιστικό Κόμμα κέρδισε με 52% των ψήφων και η Μάγια Σάντου από το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης ήρθε δεύτερη με σχεδόν 48%. Η διαφορά στις ψήφους ήταν ε, περίπου 69.000. Ο δεύτερος γύρος των εκλογών ε, ουσιαστικά έγινε σε καθεστώς ελευθερίας. Ήταν ήρεμη η μέρα των εκλογών. Η ε, συνολική καταμέτρηση των ψήφων ήταν και η απεικόνηση των ψήφων ήταν θετικό. Ακολουθήθηκαν οι διαδικασίε όπω έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν διάφορε δυσκολίε για του Μολδαβού να ψηφίσουν στο εξωτερικό. Και αυτό ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπήρξαν αναφορές ε, ότι οι Μολδαβοί πολίτες ε, έπρεπε να ταξιδέψουν ε, μακριά για να φτάσουν στο κοντινότερο εκλογικό κέντρο. Αναφέρθηκαν μεγάλες σουρές, ότι δεν υπήρχαν ψηφοδέλτια σε κάποια εκλογικά κέντρα και επομένως δεν ήταν δίκαιη η διαδικασία. Και πρέπει να υπάρξουν διδάγματα και οι αρμόδιε αρχέ θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις επιλογές και την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για να σας ενημερώσω. Ε, ψήφισαν ε, 38.000 στο εξωτερικό και ε, η Μαία Σάντου ήταν αυτή που προτιμήθηκε από τους κατοίκους στο εξωτερικό και η ανησυχία μου από, την πρώτο, από τον πρώτο γύρο ήταν ότι υπήρχε έλλειψη διαφάνειας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας και ε, ουσιαστικά ότι μπορεί να υπήρχε και χειραγώγηση από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό αφορούσε δραστηριότητες που συνδέονταν με τις εκλογές, αλλά και την ίδρυση των πολιτικών κομμάτων γενικότερα. Ε, αν χρειάζεται μεταρρύθμιση σε αυτό το τομέα και η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και προεκλογική εκστρατεία θα πρέπει να ελέγχονται αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο γύρο έγινε εμφανές ότι το νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας ε, δεν ε, θίγει αποκλειστικά το δεύτερο γύρο, δηλαδή δεν είναι σαφές αν τα όρια των δαπανών αφορούν μόνο τον πρώτο γύρο ή και τους δύο γύρους των εκλογών εγώ ζήτησα να υιοθετηθεί νομοθεσία για να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της προκλογικής εκστρατεία σε όλα τα στάδια του εκλογικού κύκλου. Ελπίζω ότι οι αρχέ στη Μολδαβία θα διερευνήσουν αυτές τις ε, ελλείψεις, τα τελήματα που εντοπίστηκαν από τους διεθνείς παρατηρητές και θα εφαρμόσουν τις συστάσεις. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή παρατήρηση των εκλογών για την επικοδομητική συνεργασία και την ομαδική δουλειά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Σόλτες. Συνάδελφο συνάδελφος Καρβινίκη, παρακαλώ, έχει το λόγο. για την Αλβανία έχουμε κλείσει αυτό το θέμα. Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι αυτά τα συμπεράσματα και συστάσεις που έκαναν οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην αποστολή είναι αντικειμενικά και κατάλληλα. Νομίζω ότι πραγματικά αντικατοπτρίζουν τι συνέβη στι εκλογέ. Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τον κύριο Σόλτε έκαναν εξαιρετική δουλειά και Πέρα από τη συμπάθεια που δείχνουμε στους εταίρους μας ε, στο Κισινάου, πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή τη φορά είχαμε και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού Φίλιπ για την διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό να πούμε ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να δείξουν ε, μια αίσθηση ευθύνη ε, όταν συζητούμε την κατάσταση στην Μολδαβία. Πρόκειται για μια χώρα η οποία έχει σκληρή ιστορία πίσω της. Δεν ε, γίνονται εύκολα δηλώσει από τους πολιτικούς. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη δημοκρατία της Μολδαβίας στο μέλλον και είναι σημαντικό η κυβέρνηση και η κοινωνία να αισθάνονται αυτή την υποστήριξη. Η κοινωνία στη Μολδαβία εξακολουθεί να είναι διαιρεμένη. Αισθάνονται οι πολίτε ότι δεν πάνε τα πράγματα προ την ορθή κατεύθυνση. Θα ήθελα επίση να καλωσορίσω μια εκδήλωση από χώρα σήμερα. Ο Πρωθυπουργό Φίλιπ επισκέφθηκε το ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και υπέγραψε μια συμφωνία να ανοίξει ένα γραφείο σύνδεσης με τον Άτομο στο Κισινάου. Και θα έλεγα ότι, <laughs> θέλω να το τονίσω αυτό, είναι γραφείο σύνδεσης και όχι στρατιωτική βάση. Ο κύριος Πρέντα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σύντομε παρατηρήσει για τι εκλογέ στη Μολδαβία. Αλλά να συγχαρώ τον κύριο Σόλτος και τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας που μετέστησαν επί τόπου. Πρώτη παρατήρηση για την προεκλογική εκστρατεία που επηρεάστηκε πολύ σοβαρά από μια ανισορροπία στη χρηματοδότηση και την επικοινωνιακή πολιτική και τη σχέση με τα ΜΜΕ. Ε, ο, δεν υπήρχε πρόσβαση για τους οπαδούς της κυρίας Μαία Σάντος στα ΜΜΕ και οι πολιτικές και διοικητικές ελίτ παρεμπόδισαν την πρόσβασή της, ε, όχι μόνο γιατί ήταν επικριτική κατά του ε, τον αλλά και του ε, συνασπισμού που ανέβηκε στην εξουσία. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αίσια διεξαγωγή των εκλογών. Οι εκλογές δεν είναι μόνο η μέρα των εκλογών. Ε, είναι αδύνατο να διανοηθείτε την έλλειψη ισορροπίας. Ε, δηλαδή δεν υπήρχαν για τη Μάια Σάντο ούτε πόστερ ούτε τίποτα. καμία διαφήμιση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, ε, σε πολλά εκλογικά κέντρα δεν υπήρχαν ε, ψηφοδέλτια. Καταλαβαίνετε πόσο κακή ήταν η οργάνωση των εκλογών. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε λοιπόν ότι εξελίχθηκαν αίσια οι εκλογές. Πότε δεν έχω ξανακούσει αυτό να έχουν τελειώσει τα ψηφοδέλτια. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι. Ε, γι' αυτό ο πρόεδρος τώρα, νέος πρόεδρος, α, έχει αναλάβει τη δέσμευση να ακυρώσει τη συμφωνία ε, σύνδεσης και ναι, ε, μετά την πίεση που δέχτηκε από διάφορους πολιτικούς παράγοντες, από διάφορα μιμιέψεων, λέει θα το σκεφτώ, ίσως όχι τελικά κτλ. Ακόμη και αν επίσημα δεν την ακυρώσει, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην εφαρμοστεί. Αν διαβάσετε το, τις προγραμματικές του δηλώσεις, ξεκάθαρα μιλάει για κατασταλτικό, απολυταρχικό καθεστώς κατά της Μολδαβίας, μιλάει για υπεριαλισμό, για ε, τον άκρατο καπιταλισμό. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι έχετε γυρίσει στη δεκαετία του 50. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε ψευδεστήσεις για αυτό το πρόεδρο ε, και ο προευρωπαϊκός προευρωπαϊκός συνασπισμός έχει αυτοανακηρυχθεί ε, σε ηγέτη αυτού του συνασπισμού. Λέγεται πλά μια Πλότικ και πρόκειται για ένα ολιγάρχη ε, δηλαδή ελέγχει αυτός ο λιγάκι στο συνασπισμό και κυβερνάται η χώρα από έναν κομμουνιστή αυτών των ντοντών. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και θα πρέπει να καταλήψουμε τις ψευδεστήσεις που έχουμε και κυρίως για κάτι μελη που έχουν άμεσα συμφέροντα ε, για τη Ρουμανία μιλάω που ε, παραμένει εγκλωβισμένη με, με αυτό που έγινε με αυτόν τον ολιγάρχη δεν ήταν ελεύθερες οι εκλογές. Να ε, επαναλάβω κλείνοντας, ε, υπήρχε δυσαναλογία σε σχέση με το χρόνο τηλεθέασης, τη διαφήμιση κτλ. Ήταν ε, που στη οργάνωση εξαιτίας ε, του κυρίου Ντοντόνα και ο νέος πρόεδρος ε, θα αντιμάχεται την Ευρώπη και ο, ο νέος συνασπισμός ελέγχεται άμεσα από έναν ολιγάρχη. Αυτή είναι η κατάσταση. Σας ευχαριστούμε. Όπως είδαμε έχουμε κάποιες παρακλίνουσες απόψεις, είναι και λογικό. Εκτός μικροφώνου η παρέμβαση είπα ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις γιατί άκουσα τον επικεφαλή της αντιπροσωπείας, άκουσα και τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας και κατόπιν άκουσα και σένα. Έχουμε διαφορετικές απόψεις, είναι λογικό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε γύρω από αυτό το θέμα της Μολδαβίας. Θέλετε κάτι να προσθέσετε ή εντάξει. Παρακαλώ. Thank Ευχαριστώ. Διαφωνώ με κάποιες από τις εκτιμήσεις του κυρίου Πρέντα και ναι, ήταν δύο υποψήφοι με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο, διαφορετική ιστορία και Μας δημιούργησε ανησυχίες όντως αυτό που είπε για τα ΜΜΕ ο κύριος Πρέντα θα είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα είναι και ευκαιρία γιατί θα συζητούμε με τον ε, νέο πρόεδρο ε, σχόλια εκτός μικροφώνου του κύριου Πρέντα. Ε, ναι, συνεχίζω, συνεχίζει ο Σόλτας, ε, είναι ο επίσημος εκπρόσωπος. Δεν γίνεται, όποιος και να είναι, όποιο και να είναι το χέρι πίσω από το συνασπισμό, αυτός ο ολιγάρχης δεν μπορούμε να, μην, να απορρίψουμε ως συνομιλητές για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ποια πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό. Ολοκληρώθηκε εδώ η συνεδρίασή μας. Το επόμενο ραντεβού στις 5 Δεκεμβρίου το απόγευμα. Σας ευχαριστώ και καλό βράδυ σε όλους.